issue. There was already a debate in the Και από πλευρά ε, τη Προεδρία και τη Κοινοβουλευτική μα Επιτροπή δίνουμε ύψιστη προτεραιότητα για αυτό το θέμα. Θα μπορούσε να καταληθεί υποχρέωση θεωρήσεων διαβατηρίων μέχρι τον Ιανουάριο 2010 η γήτρια κυρία Τάνια Φαζόν εργάστηκε έντονα τις τελευταίες εβδομάδες. Κατέθεσε την, το σχέδιο έκθεση της και το, την αποστολή για το, στο Σαράγεβο και την ε, επιτήρηση ένα από τα πιο, σημαν, πιο επίμαχα θέματα σε αυτό το χαρτοφυλάκιο. Υπό την ιδιότητά της λοιπόν ως εισηγήτρια της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών η κυρία Φαζόν θα λάβει τον λόγο πρώτη και μετά θα ακούσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Σουηδική Προεδρία τα σχετικά. Η κυρία Φαζόν παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Όπως είπατε είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα. Σε αυτό το σημείο θα περάσω στα σλοβενικά σε αυτή την πρώτη μου παρουσίαση. Θα μιλήσω τη γλώσσα μου. Σας ευχαριστώ λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι που μου δώσατε τον λόγο, εκπρόσωποι της Επιτροπής του Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι προετοίμασα το σχέδιο έκθεσης όπως ακούσατε αφού μελέτησα σε εξειδικευμένα σε βάθος της... Ε, συνθήκες στα Δυτικά Βαλκάνια και μελέτησα την προθυμία των χωρών για διευκόλυνση θεωρήσεων διαβατηρίων. Όλα αυτά υπό το φως των προσπαθειών που καταβάλλονται ότι θα έπρεπε να ολοκληρώσει τη διαδικασία απελευθέρωσης θεωρήσεων διαβατηρίων η Ευρωβουλή όσο το δυνατόν νωρίτερα. Η πρόταση που έχετε στα χέρια σας είναι κατά κάποιο τρόπο ένα συμβιβασμός που συμφωνήθηκε και έλαβε την υποστήριξη και όλων των τριών σχεδόν εισηγητών και θέλω να τους ευχαριστήσω για το έργο που επετέλεσαν τους σκιώδεις εισηγητέ. Είδαμε μια παρόμοια συζήτηση για την απελευθέρωση των θεωρήσεων διαβατηρίων στην Επιτροπή, Συνταγματικών, ε, στην Εξωτερικών Υποθέσεων, ΑΦΕΤ, εχθές. Γιατί είναι σημαντικό λοιπόν να καταργηθούν οι απαιτήσει θεωρήσεων διαβατηρίων για όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Θα ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς σήμερα ότι μόνο δύο βήματα από τη χώρα μας υπάρχουν νέες γενναίες που αποκλείονται και απομονώνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχουν δυνατότητα να ταξιδέψουν σε αυτήν. Αυτές οι γενναίες των νέων μετά τους πολέμους της Ιουγκοσλαβίας που χώρισαν τις οικογένειές τους και χώρισαν και τις χώρες τους. Ξέρουν όσα γνωρίζουν για τους Ευρωπαίους όπως όσα γνωρίζουν για τους Αμερικανούς από το διαδίκτυο. Κατανοούν το μέλλον και το μέλλον της χώρας τους και αν δεν έχουν τα δικαιώματα, θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της Ένωσης, ε, για παράδειγμα το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας, να σας υπενθυμίσω ότι σύμφωνα με την ατζέντα της ε, Θεσσαλονίκης, οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων αποκτούν ε, μια σαφέστατη προοπτική Είχαμε και σε σχέση με την ΦΥΡΟΜ το Μαυροβούνιο, να υπάρξει η δυνατότητα των χαλαρώσεων αυτών. Δεν θα απαιτείται από τον Ιανουάριο 2010 θεώρηση διαβατηρίων για αυτούς τους πολίτες αυτών των χωρών. Θα ήθελα όμως παρόλα αυτά να επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι τον Ιούλιο, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε αυτή την πρόταση, μόνο μία χώρα τότε υλοποιούσε όλες τις προϋποθέσεις ε, που είχαν τεθεί ως γνώμονα 100% γιατί δεν συμπεριέλαβε τη Βοσνία Ζεγοβίνη και την Αλβανία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της. Δεν το γνωρίζω το γιατί. Όμως η εικόνα σήμερα έχει αλλάξει, έχει μεταβληθεί. Μετά τις ε, εκθέσεις ε, που υπευλήθησαν από το Μαυροβούνιο ή από την Βοσνία, Ζεγοβίνη και Αλβανία την προηγούμενη εβδομάδα διορθώνει η ομιλήτρια μπορούμε να δούμε ότι προσεγγίζουν την υλοποίηση των, ε, υλοποιούν τα κριτήρια και αυτό θα πρέπει να το σημειώσει και να το λάβει υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σημαντική πρόοδο σημειώθηκε μετά από την δημοσιοποίηση της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επίσης και σε άλλες χώρες. Ιδιαίτερα για τη Βοσνία το γεγονός ότι δεν είχε συμπεριληφθεί στον πρώτο γύρο απελευθερώσεων από τις θεωρήσεις διαβατηρίων θα έχει σημαντικές επιπτώσεις, διότι μόνο οι Βόσνοι θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα υποστούν το πλήγμα από την ε, ε, επιβολή θεωρήσεων διαβατηρίων. Όπως ακούσατε θα, σε σχέση με την ε, αποστολή μας στο Σαράγεβο θα μπορέσω να μελετήσω επιτόπου τα σχετικά στοιχεία και θα δω αν είναι σε θέση να υλοποιήσει και τι κάνει αυτή η χώρα σε σχέση με τα κριτήρια. Ήδη μπορώ να σας πω ότι έχουν προοδεύσει και εκδίδουν βιομετρικά διαβατήρια. Τώρα για το πόσο γοργά μπορεί να τυπώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια νέα έκθεση και κατά πόσο θα ληφθεί αυτή η πρόοδος στη Βοσνία υπόψη, τώρα βρισκόμαστε στα μέσα της Υπάρχει ακόμα δυνατότητα να αλλάξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την θέση της του Ιουλίου. Η έκκλησή μου είναι απλούστατη. Ας επιτρέψουμε στη Βοσνία Ζεγοβίνη και στην Αλβανία να έχουν τη δυνατότητα να πιάσουν το τρένο με τις άλλες τρεις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, να επιβιβαστούν σε αυτό το σιδηρόδρομο και να μπορέσουν, να υλοποιήσουν όλα τα κριτήρια τα οποία έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι για να τους δώσει κανείς ε, κάποια κατεξαίρεση ε, έγκριση όταν έρχεται η ώρα υλοποίησης κριτηρίων. Είναι η δυνατότητα να μπορέσουν υπό όρους ε, να δούμε ότι θα ενταχθούν και αυτές οι χώρες με τις υπόλοιπες. Δεν θα χάσουμε χρόνο τροποποιώντας αυτόν τον κανονισμό στο μέλλον. Δεν θα χρονοβορήσουμε. Θα είναι σαφέστατο μήνυμα επίσης προς τους πολίτες αυτών των δύο χωρών. Θα γνωρίζουν ότι απευθύνουμε έκκληση στις κυβερνήσεις τους να ολοκληρώσουν το έργο των μεταρρυθμίσεων και θα ωφεληθούν οι πολίτες από τα άμεσα αποτελέσματα που θα είναι θετικά. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι έγινε πρόοδος, αλλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και τις πολύ ευαίσθητες προϋποθέσεις και συνθήκες που επικρατούν στη Βοσνία Ζεγοβίνη σήμερα και στην Αλβανία. Γι' αυτό πιστεύω, για αυτούς τους λόγους, πιστεύω ότι είναι αναγκαίο να υλοποιηθούν οι προϋποθέσεις ε, που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως κριτήρια. Όμως από την άλλη πλευρά πιστεύω επίση ότι δεν υπάρχει κανένα λόγο. Δεν υπάρχει λόγο να δημιουργούνται περαιτέρω εντάσεις σε αυτή την περιοχή, διότι ταχύτατες αποφάσεις ε, μπορεί να έχουν σοβαρές ε, επιπτώσεις. Τα Δυτικά Βαλκάνια είναι μια περιοχή που χρειάζεται τη βοήθειά μας και εμείς ε, προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε τη σταθερότητα εκεί. Ξέρω ότι υπάρχουν επικρίσεις εις βάρος της πρότασής μου από κάποιους. Λένε ότι θα μπορούσε να ερμηνευτεί ότι όλα ολοκληρώθηκαν και επετέφθησαν και θα μπορούσαν έτσι να σταματήσουν οι μεταρρυθμίσεις ίσως. Όμως εγώ είμαι πεισμένη ότι αν η Ευρωβουλή υποστηρίξει τις προτάσεις μου και πιστεύω ότι καταρχήν υπάρχει αυτή η υποστήριξη, είναι δεδομένη αυτή η υποστήριξη για τις θέσεις μου, θα στείλουμε ένα έντονο ισχυρό μήνυμα στους πολιτικούς στη Βοσνία Ζεγοβίνη επιτόπου ότι η ευθύνη είναι δική τους. Εκείνοι είναι υπεύθυνοι να συνεχίσουν το έργο για να ανοίξουν οι πύλες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση προ χάρη των πολιτών τους. Πιστεύω ότι θα μπορέσουν να υπομισθούν αυτή την ευθύνη και θα δείξουν προθυμία να ανταποκριθούν ο χρόνο έδειξε ότι έχουν προχωρήσει σημαντικά στι μεταρρυθμίσεις του τελευταίου μήνε. Υπάρχει επίση και η ιστορία του Κωσυφοπεδίου που είναι τελείω διαφορετική από τη Βοσνία Ζεγοβίνη και την Αλβανία. Στην πρότασή μου προσπαθώ σε σχέση με αυτό να δώσω μια πολιτική πρωτοβουλία, να αναλυφθεί πολιτική πρωτοβουλία. Δεν συσχετίζεται αυτό με την αναγνώριση του Κωσυφοπεδίου. 22 κράτη-μέλη έχουν αναγνωρίσει το Κωσυφοπέδιο ω οντότητα, 5 όχι. Δεν έχει κάποια σχέση ε, σε σχέση με την αναγνώριση αυτό, αλλά είναι το θέμα της ε, διευκόλυνσης ε, ε, που πρέπει να λάβουμε υπόψη όσον αφορά την ατζέντα. Παρότι υπάρχει αυτή η πολιτική κατάσταση όμως δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε τους πολίτες του Κωσυφοπεδίου σε μια μαύρη τρύπα και να αγνοηθούν εκεί, να ε, μείνουν εκεί. Πρέπει να γίνει η προσπάθεια να εξευρεθεί ένας τρόπος που θα δώσει την δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριλάβει το Κωσυφοπέδιο ή να ξεκινήσει κάποιο είδους διαπραγματεύσεις ή κάποιο είδους διάλογο με το Κωσυφοπέδιο όσον αφορά τις απελευθερώσει από την υποχρέωση για θεωρήσεις διαβατηρίου χωρίς να προδικάζουμε το τι θα γίνει τελικά με την αναγνώριση του κοσυφοπεδίου ή όχι. Και έτσι λοιπόν ε, σε παράλληλη τροχιά πρέπει να ανοίξει η πύλη της Ευρώπης και για αυτούς τους κοσοβάρους επίσης. Ευχαριστώ. John. you, ευχαριστώ κύριε Φαζιάν Τώρα ας ακούσουμε από τη Σουηδική Προεδρία τα σχετικά. Η κυρία Ιστονσον παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, όπως ε, προαναφέρθηκε, αυτή είναι μια πολύ σημαντική πρόταση και η απόφαση που πρέπει να ληφθεί για πάρα πολλούς πολίτες, για πάρα πολλούς ανθρώπους θα έχει τεράστια σημασία. Την 1η Ιανουαρίου 2008 ε, είχαμε την πρώτη συμφωνία με χώρες ε, των Δυτικών Βαλκανίων που άρχισε να ισχύει τότε και μετά κάποιους μήνες υστερότερα ξεκίνησε ο διάλογος ε, για την απελευθέρωση από τις θεωρήσεις διαβατηρίων. Ε, συγκροτήθηκε, κατατίστηκε ένα χρονοδιάγραμμα. Τρεις χώρες, η Μακεδονία, η Σερβία και το Μαυροβούνιο υλοποιούν, η Φύρομ, η Σερβία και το Μαυροβούνιο υλοποιούν τα κριτήρια ή σχεδόν τα υλοποιούν. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να τηρήσει τα υπεσχημένα η Ευρωπαϊκή Ένωση και να αρχίσει να ισχύει η απελευθέρωση θεωρήσεων διαβατηρίων για τους πολίτες αυτών των χωρών. Είναι σημαντική προτεραιότητα της Σουηδικής Προεδρίας αυτή η υπόθεση. Θέσαμε ως στόχο ενώπιον μας ότι στην συνεδρίαση του Συμβουλίου από την 30 η Νοεμβρίου στις 1η ε, Δεκεμβρίου θα πρέπει να ρυθμιστεί το θέμα ώστε από, το 2010 να απελευθερωθούν από τις θεωρήσεις διαβατηρίων οι πολίτες αυτοί. Να δώσουμε επίσης να ενθαρρύνουμε την Βοσνία Ζεγοβίνη και την Αλβανία να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους ώστε να απαλλαχθούν και αυτές οι χώρες από τις θεωρήσεις διαβατηρίων στη συνέχεια. Είναι πολύ σημαντικό να επισημάνουμε ότι η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει τερματιστεί με κανέναν τρόπο. Είναι μια ανοιχτή διαδικασία. Θα επανέλθω στο θέμα αυτό και για την χρονική απελευθέρωση αυτή. Θα πρέπει, αν θέλουμε να κάνουμε κάποιες τροποποιήσεις, θα ήταν δύσκολο να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα. Αν θέλουμε να έχουμε σημαντικές αλλαγές, τότε θα μπορούσε από δεν θα μπορούσε να τηρηθεί η ημερομηνία της 1ης Ιανουαρίου 2010 για την απελευθέρωση από διαβατηρίων. Και έτσι θα χάναμε την αξιοπιστία μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα τηρούσαμε τα υπεσχημένα. Η ελευθέρωση από διαβατηρίων πρέπει να γίνει λοιπόν όπως το σχεδιάσαμε μέσα στην προθεσμία αυτή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Τώρα θα ακούσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Γκόγκου παρακαλώ. Ε, Καλημέρα. Εγώ ήδη παρουσίασα τις ε, γενικές γραμμές της προτάσεως της Κομισιόν εχθές και θα σταθώ τώρα και στην ε, πρόταση, της, στον πολιτικό χαρακτήρα της πρότασης όπως διατυπώθηκε από τον Επίτροπο Μπαρό πριν από μερικές μέρες στο Στρασβούργο. Θα προσπαθήσω λοιπόν να διευκρινίσω μερικά πράγματα μετά από όσα άκουσα και από την Προεδρία και από τον εισηγητή. Θέλω να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για την ε, υποστήριξη που μας δίνουν όλες οι πολιτικές οικογένειες σε αυτή την πρόταση. Δηλαδή υπάρχει μία ε, βλέπουν όλες οι ομάδες με καλό μάτι αυτήν την απολευθέρωση της ε, υποχρέωσης ε, θεώρησης. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει σήμερα η συζήτηση στην έκθεση αυτή να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα από τεχνικής πλευράς. Τώρα, για τη διαδικασία αξιολόγησης Επιτρέψτε μου να επανέλθω για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Ε, δόθηκε η εντύπωση ότι υπάρχει μία χώρα που εφαρμόζει τα κριτήρια Δηλαδή η ΦΥΡΟΜ ε, πληρεί τα κριτήρια και άλλες όχι. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι σωστό. Θα πρέπει να το δούμε αυτό διαδοχικά με το πώς ε, θα προχωρήσουμε τον Ιανουάριο του το πώς προχωρήσαμε μάλλον τον Ιανουάριο του 2008 στην απολευθέρωση των θεωρήσεων από την ε, πολιτική συνεργασία της Σλοβενικής Προεδρίας και κατόπιν πρόταση της Κομισιόν. Λοιπόν, έχουμε δύο φάσεις. Οι δύο φάσεις απαιτούν καταρχήν πληροφορία γραπτός. Θέλουμε να έχουμε όλες τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για να εκπληρώσουμε το φύλλο πορείας. Στα τέλη του 2008 αποφασίστηκε επί τόπου να γίνει μία αξιολόγηση και καταβλήθηκε μία τεράστια προσπάθεια από την Κομισιόν και με υποστήριξη των εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών για να διαπιστώσουν επί τόπου ότι όντως οι μεταρρυθμίσεις εφαρμόστηκαν. Πρόκειτο λοιπόν για ένα σχέδιο πάρα πολύ σημαντικό Δηλαδή εντάξει μεταρρυθμίσεις στο χαρτί, αλλά θα πρέπει οι μεταρρυθμίσεις να γίνονται και στην πράξη. Αυτή ήταν λοιπόν η δεύτερη φάση του σχεδίου αξιολόγησης και είχαμε την έκθεση του Μαΐου της Κομισιόν και μετά την πρόταση της Κομισιόν για την απολευθέρωση των θεωρήσεων ε, για την ε, Σερβία, το Μαυροβούνιο και τη Φύρομ. Γιατί θεωρήσαμε δηλαδή ότι αυτές οι χώρες είχαν τη δυνατότητα να εκπληρώσουν όλα τα κριτήρια. Και ορίσαμε εμείς την πρόταση της Κομισιόν ποια σημεία θα πρέπει να επαληθεύσουμε. Το είπα και χθες ότι για το Μαυροβούνιο και για τη Σερβία έχουμε κάνει τις αποστολές στο παρελθόν, επαληθεύσαμε τι έπρεπε να επαληθεύσουμε, αλλά και τον επόμενο μήνα θα ξαναπάμε για να δούμε τα τελευταία που μένουν. Αυτό είναι και το πλαίσιο αξιολόγησης. Όταν υπέβαλε αυτές τις προτάσεις η Κομισιόν για αυτές τις χώρες, το είχε καθαρό ότι θα γινόντουσαν αποδεκτοί όλοι οι όροι μετά από την έγκριση τον Ιούλιο. Και οι όροι αυτοί θα άρχισαν να ισχύουν μετά από μερικές εβδομάδες. Τώρα πάμε στην Αλβανία και στη Βοσνία. Διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν σημαντικές πρόοδοι υπήρχε μία συνέργεια με αυτές τις χώρες, τεράστια συνέργεια και κατάφεραν ε, τεράστιες ε, ε, πρόοδους. Μεγάλες μεταρρυθμίσεις οι οποίες εφαρμόστηκαν. Όμως την αξιολόγηση που έγινε διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν ακόμη ουσιαστικότατα σημεία τα οποία θα πρέπει να διορθωθούν. Όχι μόνο το θέμα των διαβατηρίων και στα τέσσερα μπλοκ έχουμε, έχω εδώ καταλόγους και καταλόγους με σημεία που πρέπει να, ε, να εκπληρωθούν. Ας πούμε το θέμα των μεταφορών. και στην έκδοση των διαβατηρίων. Γιατί εμείς ε, σήμερα απαιτούμε βιομετρικά διαβατήρια. Και δεν το απαιτούμε μόνο σε αυτούς και στους δικούς μας τους πολίτες το απαιτούμε. Περιμένουμε λοιπόν τώρα για την Αλβανία αρχές Οκτωβρίου την επίσημη αξιολόγηση. Εμείς είπαμε, αξιολογήσαμε επί χάρτου πρώτα το τι έγινε και ξεκίνησαν αποστολές αξιολόγησης οι οποίες μέχρι τα τέλη του χρόνου θα ολοκληρωθούν ως, με το συγκεκριμένο πρόγραμμα για να δούμε και επί τόπου τι κάνουν οι Αλβανοί με τις μεταρρυθμίσεις Ο Αντιπρόεδρος Μπαρό ήδη εξήγηλε στο Στρασβούργο την πρόθεση της Κομισιόν να παρακολουθήσει από κοντά όλη αυτή τη διαδικασία και να υποβάλει προτάσεις ε, εάν το 2010 αν εκπληρωθούν όλα τα κριτήρια. Ένα σχόλιο το αρδικό μου εγώ εχθές αναφέρθηκα σε αυτά τα οποία προτείνει το Κοινοβούλιο για την πραγματική κατάργηση του καθεστώτος της ε, βίζας ε, για την Βοσνία και για την Αλβανία. Και με αυτή την πρόταση τέλος πάντων, με αυτή την προσέγγιση αστερίσκων θέλετε, εγώ είμαι έτοιμη να σας εξηγήσω αναλυτικότερα όλη αυτή την πλευρά του αστερίσκου δηλαδή που ανέφερα και να σας πω το τι σκεφτόμαστε εμείς στην Κομισιόν γι' αυτό. Η Κομισιόν ανέφερε σαφώς την πρόθεση της να εκπονήσει μία μελέτη και να δει πώς θα προχωρήσουμε με μία πρόταση φτιαγμένη στα μέτρα της κατάστασης αυτής της χώρας. Και αυτό μέσα στο πνεύμα το οποίο διέπει γενικώ τις σχέσεις μας με τα Δυτικά Βαλκάνια. Αλλά πρώτα θα πρέπει να εφαρμόσουμε τις ε, συμφωνίες διευκόλυνσης και θέλουμε επίσης να έχουμε και εγγύησεις, να δούμε ποιος θα είναι ο εγγυητής ούτως ώστε να έχουμε συγκεκριμένες εγγύσεις ποιος θα είναι υπεύθυνο σε περίπτωση επανεισδοχής, κυρίως από τις αρχές του κοσυφοπεδίου. Σας ευχαριστούμε. Πολλοί ευρωβουλευτές έχουν ήδη ζητήσει το λόγο για το ζήτημα αυτό. Να σας πενθυμίσω όμως ότι ε, βρισκόμαστε στο σημείο 17 της ημερήσιας διάταξης. Έχουμε πολλά σημεία να καλύψουμε μέχρι το 34 που θα πρέπει να καλύψουμε δηλαδή σήμερα. Σας παρακαλώ λοιπόν πολύ να το έχετε αυτό κατά νου κάθε φορά που παίρνετε το λόγο και να είστε σύντομοι στις παρεμβάσεις σας. Να κάνετε δηλαδή μια καλή χρήση του χρόνου. Μιλήστε μέγιστο δύο λεπτά, παρακαλώ πολύ, ο καθένας. Ο κύριος Μπουζουτήλ έχει πρώτο το λόγο, παρακαλώ. Οι σκιώδεις μάλλον εισηγητές πρώτα. Κρατσαβίλτ πρώτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να σας πω ότι ε, εκτίμησε ιδιαίτερα τη συνεργασία με την κυρία Φαζόν και την Σάρα Λούτφορντ και χαίρομαι πάρα πολύ που πολλές από τις παρατηρήσεις που βάλαμε εμείς ως ΕΛΚ έχουν συμπεριληφθεί στην τελική τώρα έκθεση. Είναι πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό το ότι συμφωνούμε ότι θα πρέπει να καταβληθούν όλες οι προσπάθειες προκειμένου να επιταχυθεί η διαδικασία απελευθέρωσης υποχρέωσης θεώρησης για όλους τους λαούς των Δυτικών Βαλκανίων. Θα πρέπει να ζητήσουμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμόσει την, την απόφαση Συμβουλίου μόλις αυτή υιοθετηθεί. Και δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε εδώ πέρα προβλήματα όσον αφορά τα κριτήρια, δηλαδή να σεβαστούμε τα κριτήρια αυτά. Το ΕΛΚ ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τους ανθρώπους αυτούς, για τη νέα αυτή γενιά ανθρώπων που αισθάνονται ουσιαστικά μπλοκαρισμένοι στην περιοχή αυτή. Κανείς, σε καμία περίοδο, στην, κανείς από την περιοχή αυτή δεν θα πρέπει να μην μπορεί να κυκλοφορήσει ελεύθερα. Θα πρέπει να προωθήσουμε μια ρεαλιστική άποψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά ας μην προσπαθούμε εδώ πέρα να κοροϊδέψουμε τους ανθρώπους της Βοσνίας στο σημείο 6 για παράδειγμα που χρησιμοποιείτε τους αστερίσκους για τη μεταφορά από τον αρνητικό στο θετικό κατάλογο στην πραγματικότητα τα πράγματα δεν διευκολύνονται για την Βοσνία. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό το πράγμα Τάνια από το να θέτει κανείς προϋποθέσεις και κίνητρα είναι ένα πολύ σημαντικό πολιτικό κίνητρο από μόνο του. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δώσουμε τη δυνατότητα στις ε, αρχές της Βοσνίας να κινηθούν προς την κατάργηση υποχρέωσης θεώρησης και έχουν καταβάλει φοβερές προσπάθειες μέχρι στιγμής. Για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή να προχωρήσουμε με ένα διαφορετικό τρόπο και να καθυστερήσουμε τελικά την όλη διαδικασία κατάργηση υποχρέωσης θεώρησης και για τους ε, Βόσνιους. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε μια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον, την Άνοιξη και να ανοίξουν τα σύνορα το καλοκαίρι. Για ποιο λόγο λοιπόν να χρησιμοποιούμε τον αστερίσκο αυτή τη στιγμή, για ποιο λόγο να κρύβουμε τα κριτήριά μας. Εμείς ενδιαφερόμαστε για όλους τους λαούς των Δυτικών Βαλκανίων, είτε είναι Σέρβοι, είτε είναι Αλβανοί, είτε είναι Βόσνοι είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι είμαστε ανοιχτοί για περαιτέρω διάλογο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε, κυρία Λούτφορντ. Uh, Μπορώ να πω ότι μου δημιουργήθηκε κάποια σύγχυση με αυτά τα οποία άκουσα. Εγώ είμαι συντάκτρια γνωμοδότησης για την Επιτροπή ΑΦΕΤ. Δεν είχα καταλάβει ότι η κυρία Κρατσαμπίλτερ αυτή τη στιγμή ουσιαστικά αποχωρεί, απομακρύνεται από την κοινή θέση που είχαν αποφασίσει όλοι οι σκιώδεις ηγητές. Και χθε στην ΑΦΕΤ υπήρχε γενική υποστήριξη για το σύστημα το οποίο προβλέπεται εδώ πέρα με μια λίγο διαφορετική διατύπωση. κύριος Πόσολτ, την κυρία Πάκα από το ΕΛΚ και άλλοι συναδέλφοι από το ΕΛΚ θέλουν να συμπεριλάβουν και τις πέντε χώρες στα πλαίσια του πεδίου εφαρμογή του υφιστάμενου κανονισμού, το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό από το να έχουμε τώρα έναν κανονισμό και έναν διαφορετικό κανονισμό στο μέλλον. Ελπίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Κανείς δεν θέλει να υποβαθμίσει τα κριτήρια και νομίζω ότι αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στην έκθεση τη κυρία Φαζόν. Δεν θέλουμε να υποτιμήσουμε σε καμία περίπτωση συμβολή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής επίσης και γι' αυτό το λόγο η διάρθρωση τη επιτροπή τη κυρία Φαζόν, η δομή που ακολουθεί η έκθεση αυτή, είναι ότι θα πρέπει όλοι να συμπεριλαμβάνονται στην, στο πεδίο εφαρμογή, αλλά η εφαρμογή του Visa Waiver για τη Βοσνία, Ερζεγοβίνη και την Αλβανία εξαρτώνται από την αξιολόγηση που θα κάνει πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και από ό,τι κατάλαβα θα γίνει για τις δύο αυτές χώρες η αξιολόγηση πριν τα τέλη του έτους και η αξιολόγηση αυτή ενδεχομένως να οδηγήσει, να μην οδηγήσει τελικά σε μια ταχεία διεκπαιρέωση της κατάστασης και των χωρών αυτών όσον αφορά δηλαδή την κατάργηση υποχρέωσης θεώρησης. Αυτό που έχει σημασία και αυτό που μετράει, ανεξάρτητα από, οτιδή, από οτιδήποτε άλλο υπόθηκε αυτή τη στιγμή, είναι η αξιολόγηση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή θα καθορίσει τελικά αν αυτέ οι δύο χώρε οι οποίε αναφέρθηκα θα περάσουν στον τελικό κατάλογο. Όσον αφορά τώρα του αστερίσκου που χρησιμοποιούνται στι τροπολογίε, νομίζω ότι και αυτό θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε ενδεχομένω λίγο αργότερα στη συζήτηση που θα γίνει. Δεν κατάλαβα πάντω, ακούγοντα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Συμβούλιο, ποια είναι η βασική του αντίρρηση στα όσα προτείνονται όσον αφορά δηλαδή την Βοσνία και την Αλβανία. Από ό,τι φαίνεται υπάρχουν προβλήματα πρακτική και νομική φύση. Δεν μπορώ να καταλάβω όμω ποια είναι τα προβλήματα αυτά. Η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη ίσχυε για δύο επίπεδα. Έλεγε δηλαδή ότι η ΦΥΡΟΜ έχει πληρώσει τα κριτήρια και ότι θέλουμε και η Βοσνία να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο και ότι αυτό θα γινόταν μέχρι τον Νοέμβριο. Ποια είναι η βασική αντίρρηση λοιπόν να ακολουθήσουν μια διαδικασία, μια δομή σε τρία επίπεδα για την εφαρμογή του κανονισμού αυτού. Και μου έκανε εντύπωση η παρέμβαση της Προεδρίας, που από ό,τι φαίνεται υπονοεί ότι η δική μας προσέγγιση, το Κοινοβουλίο δηλαδή, σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα καταφέρει να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα για τον ε, ε, Ιανουάριο για το visa waiver όλων αυτών των χωρών. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο λέγεται κάτι τέτοιο από την Προεδρία. Είναι ουσιαστικά σαν να προσπαθούν να μας εκβιάσουν. Σαν είμαστε εμεί τελικά οι υπεύθυνοι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την επιβράδυση διαδικασία για τις τρει τρεις χώρες που αναπομένουν στον κατάλογο. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο λέγεται αυτό από την Προεδρία και για ποιο λόγο παρουσιάζεται σαν μια απειλή. Νομίζω ότι γι' αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε κάποιες θεωρητικές υποσχέσεις. Το σημαντικό είναι να δούμε τι κάνουν οι εθνικές αρχές στην Βοσνία και στην Αλβανία. Το σημαντικό είναι να ισχύει η αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία θα λειτουργήσει τελικά σαν κίνητρο για τις εθνικές αρχές των χωρών αυτών, προκειμένου δηλαδή να αρχίσουν να εφαρμόζουν τα κριτήρια και τις δικές μας προποθέσεις το ταχύτερο δυνατό. Ευχαριστώ. Η κυρία Ernst, παρακαλώ. Φαίνεται ότι... Διαδικαστικό εσείς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω θα ήταν χρήσιμο αν μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας εξηγήσει για να αποσαφηνίσει ίσως προς την κυρία Λάνφορντ τις επιπτώσεις του αστερίσκου, τις πρακτικές και νομικές επιπτώσεις που απορρέουν από αυτό. The Commission η Επιτροπή παρακαλώ για την αποσαφήνιση, αλλά σύντομα παρακαλώ, σύντομα. Euh, Θα είμαι πανσύντομη. Πραγματικά μας κολακεύει η εμπιστοσύνη του Κοινοβουλίου. Εμείς όλη αυτή τη διεργασία την κάνουμε με τη βοήθεια των εμπειρογνωμόνων, ε, που μας παρέχουν τα κράτη-μέλη για να κάνουμε όλη αυτή τη δουλειά. Σύμφωνα με την έκθεση του Κοινοβουλίου, το Κοινοβούλιο προτείνει να λάβουμε μία απόφαση τώρα για τις πέντε χώρες και για δύο χώρες να αναστείλουμε και αυτό μετά από την ε, δημοσίευση της έκθεσης της Κομισιόν. η Κομισιόν είναι έτοιμη να την κάνει αυτή την έκθεση. Αλλά αυτή η έκθεση θα πρέπει να συζητηθεί. Και θα πρέπει τα συμπεράσματα της ε, έκθεσης ε, της ε, Κομισιόν πρέπει να τη συμμερίζονται και τα κράτη-μέλη. Δεν μπορούμε εμείς με μία ανακοίνωση να υποκαταστήσουμε μία απόφαση που έχει ληφθεί με το Συμβούλιο. Εσείς βλέπετε την Κομισιό να λέει πολύ ωραία, πολύ σωστή αξιολόγηση για την Αλβανία και το φαντάζεστε δηλαδή ότι αύριο στα καλά του καθομένου θα αναστείλουμε την θεωρήσεις για την Αλβανία και θα κλείσουμε τα προξενία. Μα η Κομισιόν δεν διαχειρίζεται τις προξενικές αρχές, τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα και η διαχείριση, όλη, αυτή η διαχείριση σημαίνει ότι και το Συμβούλιο πλέον ε, συμμετέχει ενεργά στη λήψη της απόφασης, είναι αυτό που αποφασίζει. Τι έγινε για τη Ρουμανία, με τη Ρουμανία το 2001. Η Κομισιόν είχε παρουσιάσει μία έκθεση, πολύ λιγότερο αναλυτική με την έκθεση που παρουσιάζουμε σήμερα. Και μετά έγινε συζήτηση, μακροσκελέστατη συζήτηση στο Συμβούλιο. Και μετά από αυτό έγινε, λήφθη μία πολιτική απόφαση του Συμβουλίου, ένας νέος κανονισμός του Συμβουλίου που πρόβλεπε την κατάργηση του αστερίσκου. Αν καταλαβαίνω τώρα την πρόταση του εισηγητή, δεν θέλει να υπάρξει μία επόμενη ε, πολιτική απόφαση αλλά οι πολιτικές επιπτώσεις των αποφάσεων της Κομισιόν δεν ορίζονται από την ίδια. Δηλαδή δεν είναι η Κομισιόν εκείνη η οποία θα πρέπει να ορίσει πότε σταματάμε να απαιτούμε θεώρηση και πότε θα κλείσουμε τα προξενία. Εσείς για δύο λεπτά. Εντάξει. Δεν καταλαβαίνω απόλυτα, πρέπει να πω ειλικρινά, τις επι, ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι οι προτάσεις της κυρίας Φαγιόν, όπως εμπεριέχονται εδώ, αποσαφηνίζουν προοπτικές. Δεν είναι τεχνικό ζήτημα το οποίο συζητούμε εδώ. Είναι βαθιά πολιτικό ζήτημα, εντάξει, ότι σε αυτή την περιοχή, σε αυτή την περιφέρεια που αυτές οι πέντε χώρες έχουν μια παλαιότερη ιστορία, μια προϊστορία, το σημαντικό είναι τα κοινά στοιχεία να προαγάγουν, να προωθήσουν και γι' αυτό είναι σημαντικό να υπάρξουν τοποθετήσεις και για την Βοσνία Ζεγοβίνη και φυσικά και για το Πέδιο και νομίζω αυτές οι τοποθετήσεις αφήνουν, πρέπει να αφήνουν περιθώριο εκείνα που πρέπει να γίνουν και να επιτευχθούν σε αυτές τις χώρες ώστε να ανταποκριθούν στα benchmarkings, δηλαδή στις προδιαγραφές και στις ε, όρους, όρους και προϋποθέσεις να μπορέσουν να προωθηθούν. Υποστηρίζω αυτή την πρόταση. Τα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν τα κατανοώ. Δεν κατανόησα την δική της παρέμβαση επ' αυτού. Μία σκέψη να εκθέσω. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το κοσυφοπέδιο να κατοχυρωθεί έτσι εδώ και να διατυπωθεί μια προοπτική γι' αυτό. Δηλαδή να εκφραστεί βούληση που θα εκφράζεται με σαφήνεια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Είναι σημαντικό αυτό για την εξέλιξη, περαιτέρω εξέλιξη της χώρας. Και για όλους αυτούς που έχουν προβλήματα τώρα εδώ, η διατύπωση εμπεριέχεται που αφορά που δεν αφορά, με συγχωρείτε, το καθεστώ του Κωσυφοπεδίου. Και αυτό εντάξει, βαίνει καλώς. Και εμεί θα είχαμε κάποια πράγματα να αναφέρουμε πώ βλέπουμε το θέμα τη αναγνώριση του Κωσυφοπεδίου. Αλλά είναι πολιτικά σημαντικό αυτό το θέμα. Δεν είναι τεχνικό ζήτημα και να έχει τεχνική σημασία. Πρέπει για τι χώρε αυτή τη περιοχή να, να υπάρξει η προοπτική μια περαιτέρω προώθηση και επίλυση των προβλημάτων. Μια, α το πω έτσι, πρόοδο που θα αποσαφηνίζεται. Ευχαριστώ. Thank you. Now, Mr ευχαριστώ. παρακαλώ, Αν δεν απαιτούνται πλέον θεωρήσεις από τις χώρες αυτές, τι είδους ελέγχο, έλεγχος θα γίνεται κάθε φορά που οι πολίτες αυτοί ταξιδεύουν εκτός από την, ε, χώρα τους και επιστρέφουν στη συνέχεια στη χώρα τους. Νομίζω ότι το σύστημα της θεώρησης ακριβώς εξασφάλιζε τον έλεγχο αυτό και απέφευγε επίσης το πρόβλημα της μετανάστευσης από τρίτες χώρες. Οι άνθρωποι οι ε, οποίοι θα ταξιδεύουν πλέον ε, με το νέο αυτό σύστημα μπορούν ενδεχομένως να δουλεύουν παράνομα σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και αν δεν έχουν βέβαια τη δυνατότητα να δουλεύουν νόμιμα. Ε, ενδεχομένως λοιπόν να καταλήξουν στην μαύρη αγορά και να πέσουν και θύματα της χειρότερης δυνατής εκμετάλλευσης, αυτή την οποία συζητήσαμε χθε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπουζουτήλ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Αναφίβολα η Επιτροπή μας δίνει πολύ μεγάλη πολιτική σημασία στην διαδικασία κατάργηση υποχρέωσης θεώρησης για όλες αυτές τις χώρες. Άκουσα τις τελευταίες αυτές εξηγήσει της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πιστεύω ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να εφαρμοστεί η πρόταση της εισηγήτριας και αυτό φάνηκε ξεκάθαρα από τις εξηγήσει που μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι θα πρέπει να βασιστούμε περισσότερο στα όσα μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό δεν υπονομεύει σε καμία περίπτωση την πολιτική σημασία που δίνουμε εμείς στο χαρτοφυλάκιο αυτό. Και συμφωνώ με την κυρία Κοράτσα Μπίλτ όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Η συγκήτρα μας λέει, ωραία, τις χώρες αυτές μπορούμε να τις βάλουμε στο θετικό κατάλογο, δηλαδή δεν θα υπάρχει υποχρέωση θεώρησης, αλλά τελικά χρειάζονται ακόμα θεώρηση, αυτό λέμε και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι σαν να μιλάμε τη γλώσσα του George Orwell από το 1984. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει εμείς να δίνουμε αυτό το μήνυμα προς τις χώρες αυτές. Είναι σαν να τους κορυδεύουμε. Τους λέμε μπέντε στον κατάλογο που δεν απαιτείται θεώρηση, αλλά τελικά απαιτείται για σας θεώρηση. Είναι αυτό λύση. Νομίζω ότι μια τέτοια λύση θα μπορούσε ουσιαστικά να γυρίσει μπούμερανγκ εναντίον μας. Και υπό το φως των πολύ ξεκάθαρων εξηγήσεων που μα έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να επανακτιμήσουμε ενδεχομένω την τοποθέτησή μα. Ενδεχομένω θα πρέπει να με άκουγε και η κυρία Φαγιόν πιο προσεκτικά. Λέω λοιπόν ότι θα πρέπει να επανεκτιμήσουμε την τοποθέτησή μα και να βρούμε μια εναλλακτική οδό. Δεν έχουμε αποκλείσει μια εναλλακτική λύση, άλλωστε έτσι δεν είναι. Η προσέγγιση που υιοθετούμε αυτή τη στιγμή μου φαίνεται και μετά από αυτά που είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν θα μπορούσε στην πράξη να εφαρμοστεί. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπόντς παρακαλώ. Το κόμμα Ελευθερία είναι κατά τη κατάργηση τη θεώρηση τη υποχρέωση θεώρηση των διαβατηρίων για τα Δυτικά Βαλκάνια. Να εξηγήσω γιατί. Όταν η Σερβία, η Φύρον, το Μοντενέγκρο βλέπουμε έχουν μεγάλο ποσοστό εγκληματικότητα, οργανωμένο έγκλημα και τεράστια διαφθορά. Δεν μάθαμε τίποτα από την ένταξη της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Διερωτώ με. Τι συμβαίνει εδώ. Είναι το πρώτο βήμα αυτό, αυτές οι χώρες κάποτε μακροπρόθεσμα να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι κάθετα ενάντιος εγώ, Είμαι, διαφωνώ απόλυτα με αυτό. Και για τη Βοσνία, Αλβανία, είμαι απόλυτα εναντίον να είμαστε υπέρ της ένταξής τους. Να σας εξηγήσω γιατί. Ας δούμε τι γίνεται στη Βοσνία. Ο ηγέτης των Βόσνιων μουσουλμάνων θέλουν, θέλει να υπάρξει κατοχήρωση εγγύηση της Σαρία του Ιερού Νόμου του Κορανίου στο Σύνταγμα της Βοσνίας. Είμαι απόλυτα εναντίον. Επιπλέον η Βοσνία είναι ασφαλής λιμένας ε, μουσουλμάνων τρομοκρατών. Είναι λιμένας στον οποίο βρίσκουν καταφύγιο οι μουσουλμάνοι τρομοκράτες. Επιτέλους θα σταματήσουμε τις ανοησίες για απελευθέρωση αποθεωρήσεις διαβατηρίων για αυτές τις χώρες. Ας μην είμαστε ανόητοι. Ο κύριος Γκάντς παρακαλώ.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 bosznia hercegovina kimarad most ebben a Φυσικά σε αυτή την περιοχή υπάρχει ένταση. Αν σε αυτή την περιοχή λείπει, λείπουν τα κίνητρα σε σχέση με την απαλλαγή από αποθεωρήσεις διαβατηρίων, τότε θα ενταθεί αυτή η ένταση. Και κάποιοι θα έχουν απαλλαγή, κάποιοι άλλοι όχι. Και ένα μέρος, θα, κάποιας, μια χώρα θα αποκλείεται από αυτή την ε, απαλλαγή. Είναι κάτι πολιτικό και δεν πρέπει να ε, αγνοήσουμε την πολιτική ευθύνη που πρέπει να υπομισθούμε και πρέπει να τονίσουμε το δυνατόν ταχύτερα να υλοποιηθούν όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις ώστε αυτές οι χώρες να μπορέσουν να υλοποιήσουν τις προϋποθέσεις απαλλαγής θεωρήσεων διαβατηρίων. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Κέλλερ παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Δεν κατανόησα πάρα πολύ καλά την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι οι αστερίσκοι σε σχέση με τις τροπολογίες ε, του Κοινοβουλίου ή την θέση της κυρίας Φαγιών δεν θέτουν κάποια ημερομηνία για το πότε θα πρέπει αυτό να ισχύει. Θέτουν απλώς όρο, η προϋπόθεση. Δεν βλέπουμε λοιπόν πώς αυτό θα καθυστερούσε και οι ε, αστερίσκοι θα άλλαζαν την ε, διαδικασία. Τώρα, κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα. Θα θέλαμε να γνωρίζουμε εμείς γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι τόσο κάθετα εναντίον αυτής της πρότασης να συμπεριληφθούν και οι πέντε, όλες οι πέντε χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Μια και η Φύρομ είναι η μόνη χώρα στα Δυτικά Βαλκάνια που υλοποιεί τις προϋποθέσεις και τους όρους και δεν κατανοούμε γιατί διαφοροποιούνται μεταξύ, Βοσνία, ε, μεταξύ Σερβίας, ε, Μαυροβουνίου, Βοσνίας, Εζεγοβίνης, Αλβανίας. Δεν το κατανοούμε. Μέχρι σήμερα, μέχρι τώρα δεν μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Το δεύτερο ερώτημα είναι, το δεύτερο ζήτημα, ποια είναι τα ακριβή αποτελέσματα, οι ακριβείς επιπτώσεις αυτής της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χωρίς τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου της κυρίας Φαγιόν για το κοσυφοπαίδιο. Τι γίνεται λοιπόν για το κοσυφοπαίδιο, πώς θα αντιμετωπιστεί, ποιες επιπτώσεις θα υπάρχουν στο κοσυφοπαίδιο και τι θα γίνει με το κοσυφοπαίδιο. Αυτό θα θέλαμε να μάθουμε. Σας ευχαριστώ. Κύριε Σόγκορ παρακαλώ. Δεν θέλετε να παρέμβετε. Ωραία. Νομίζω λοιπόν ότι Πρέπει τώρα να ακούσουμε την αντίδραση από πλευρά τη ηγήτρια κυρία Φάγιον. Α, διέτε μέρα παρακαλώ. Σα ευχαριστώ πρόεδρε. Απλά και μόνο πρόεδρε ζητώ τον λόγο να εκφράσω μια επιφύλαξη. Φοβούμαι ότι στην ισπανική αντιπροσωπεία όσον αφορά το ΕΛΚ δεν θα μπορέσουμε να δεχτούμε την τροπολογία αυτή που αφορά το κοσυφοπαίδιο υπό τους όρους στους οποίους έχει διατυπωθεί. Ευχαριστώ. Thank you. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Τώρα να ακούσουμε την τοποθέτηση της ε, ε, εισηγήτριας κυρίας Φαγιών, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ για όλες τις παρεμβάσεις σα, προτάσεις ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και όλους τους Ευρωβουλευτές μέλη τη Επιτροπής μας, συναδέλφου. Να πω για άλλη μια φορά ότι είναι πολιτική δική μας ευθύνη, πολιτική ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποστείλει ένα θετικό, δυνατό, ισχυρό πολιτικό μήνυμα σε όλε τι χώρε των Δυτικών Βαλκανίων Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη βλέποντας ότι υπάρχει ουσιαστικά συνολική συμφωνία ότι πρέπει να επιταχύνουμε τη διαδικασία απελευθέρωσης θεωρήσεων διαβατηρίων για όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλτικανίων Εκεί που βλέπω να υπάρχει κάποια διαφωνία και κάπως εκπλήσωμαι πρέπει επίσης να πω ότι ο Σκιώδης εισηγητές του ΕΛΚ σήμερα διαφωνεί με αυτά τα οποία συζητήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα όσον αφορά τον αστερίσκο για τη Βοσνία και την Αλβανία. Πρέπει λοιπόν να πω ότι διαβουλευτήκαμε και με οι δήμονες ε, νομομαθείς όταν συντάσαμε την ε, έκθεση και μπορούμε να τους ξαναρωτήσουμε να δούμε ποια είναι η άποψή τους. Άκουσα τις επεξηγήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν είμαι βέβαια ότι κατανοώ τις επιφυλάξεις και δεν είναι βέβαιο το τι θα συνέβαινε με την ε, διατήρηση ή όχι των αστερίσκων. Μπορούμε να ρωτήσουμε τους νομομαθείς ε, να βρούμε μια καλύτερη νομοθετική, αν θέλετε τεχνική, για να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτών των δύο χωρών. Μπορούμε να το κάνουμε και σε συνεργασία με τους νομομαθείς ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου για να επιληθεί το πρόβλημα επαρκώς. Για το ερώτημα του συναδέλφου ή τη συναδέλφου που διατυπώθηκε. Πρέπει να πω ότι εκπλήσωμε. Αυτό δεν είναι κάτι το καινούριο αυτό που κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ τώρα. Έτσι δεν είναι. Ουσιαστικά ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει, με άλλα λόγια, ότι δεν προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν αστερίσκους, λέει από το 2001 αν δεν κάνω λάθος σε σχέση με τον θετικό κατάλογο όταν έγιναν προτάσεις για τη Ρουμανία. Όμως από την άλλη πλευρά έκαναν μία εξαίρεση πριν από τρία χρόνια Τώρα ε, από πλευρά ε, ε, εισήγηση εγκατέλειψαν την αίθουσα. Τώρα σε σχέση με νωρίτερα να μπορούν να ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορώ να φανταστώ ότι θα μπορούσαμε να βρούμε μια λύση αν συνεργαστούμε στενά. Είμαι πρόθυμη να έχω στενή συνεργασία, να έχουμε στενή συνεργασία με νομομαθεί και σε σχέση με το Ευρωκοινοβούλιο και με, να δούμε τι γίνεται με άλλου συναδέλφου, τον κύριο Σβόμποντα για παράδειγμα. Για το Κωσυφοπέδιο θα ήθελα να τονίσω για άλλη μια φορά εδώ κάτι, ότι η τροπολογία που προτείνουμε εμείς είναι ουσιαστικά μόνο η πολιτική πρωτοβουλία που πρέπει να αναλυφθεί, να βρούμε έναν τρόπο να εντάξουμε το κοσυφοπαίδιο στη διαδικασία απελευθέρωση θεωρήσεων διαβατηρίων, χωρί να προδικάσουμε τι θα γίνει με την αναγνώριση του κοσυφοπαίδιου και το καθεστώ του και το τι συμβαίνει σχετικά Έχω μια αίσθηση που έχω αποκομίσει ότι καταρχήν στις πολιτικές ομάδες συμφωνούμε επ' αυτόν. Ευχαριστώ. Η κυρία Κοράτσα Μπίλτ παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ Τάνια Φαγιόν. Θέλω απλά και μόνο να πω ότι πραγματικά έχουμε, συμφωνώ, σημαντική πολιτική ευθύνη, ιδιαίτερα για αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή εκεί στα Δυτικά Βαλκάνια, σε αυτή την περιοχή και όπως είπε συνάδελφος πιο πριν, έχουμε και το θέμα της, ε, του να μην εξαπατήσουμε τους Βόσνιους. Έχουμε ευθύνη να είμαστε τίμοι έντιμοι απέναντί τους και παρακαλώ, δώστε προσοχή να ολοκληρώσω. Έχουμε μια πάρα πολύ ε, μεγάλη πολιτική ευθύνη. Να συνεχίσουμε να λέμε στι αρχέ των Βοσνίων, κάντε τη δουλειά σα σωστά, να θέσετε εντάξει τα του οίκου σας. Καλοχαιρετίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση του πολίτε σα. Όμω οι όροι και οι προποθέσει πρέπει να είναι σαφεί και απροκάλυπτοι. Δεν πρέπει να τους αποκρύπτουμε ή να του παρασιωπούμε. Αυτή είναι η ευθύνη μα Πρέπει να είμαστε έντιμοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Λάτφορντ. Κάποια σχόλια. Κοιτάξτε, πώς καταλαβαίνω εγώ τους αστερίσκους. Το λέει άλλωστε και το ίδιο το κείμενο. Συγγνώμη, κοιτάω την εκδοχή από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Πάντως νομίζω ότι έχει να κάνει μόνο με το ότι η εξαίρεση από την κατάργηση υποχρέωση θεώρησης ισχύει μόνο για τα διαβατήρια τα οποία είναι βιομετρικά. Πρόκειται για individual conditionality, το state conditionality βρίσκεται στο ίδιο το κείμενο του κανονισμού. Στα εκτιμώντας, στην αιτιολογική σκέψη, όπου λέγεται ότι μόνο η αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μπορούσε να οδηγήσει μετάβαση κρατών από τον ένα κατάλογο στον άλλον, από τη μία κατηγορία στην άλλη. Δεν θα πρέπει λοιπόν να συγχαίουμε τα πράγματα όσον αφορά τους αστερίσκους. Θα ήθελα πάντως να ζητήσω από την κυρία Κοράτσα Μπίλτ να ξεκαθαρίσει κάπως τα πράγματα στη συνάντηση που θα έχουμε με τους ισχυώδεις συγητές. Επίσης στην Επιτροπή ΑΦΕΤ χρησιμοποιούμε μια διαφορετική διατύπωση για το κοσφοπέδιο. Νομίζω ότι θα πρέπει εδώ πέρα να έχουμε μια τέτοια διατύπωση για το κοσφοπέδιο, όπου θα αντικατοπτρίζεται σωστά η κατάσταση, όπου θα μπορούμε ουσιαστικά να έχουμε και τις χώρες εκείνες που δεν έχουν αναγνωρίσει το κοσυφοπαίδιο και όπου θα καταφέρουμε να έχουμε τελικά μια ρεαλιστική προσέγγιση για τη χώρα αυτή. Μικροφωνισμός, δεν μπορούν οι διερμηνείς να ακούσουν. Νομίζω ότι έχει δίκιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν λέει ότι θα πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία διευκόλυνση όσον αφορά για την υποχρέωση θεώρησης. Θα πρέπει να ξεκινήσουν καταρχάς συζητήσεις όσον αφορά την ε, εισδοχή και τη διευκόλυνση για τις θεωρήσεις και στη συνέχεια να περάσουμε στο ζήτημα της κατάργησης. Θα πρέπει να καταφέρουμε, και σίγουρα αυτό δεν είναι εύκολο, να βρούμε μία δομή και μία διατύπωση, η οποία να στέκει από νομική πλευρά και να αντικατοπτρίζει τελικά τα πιστεύω που έχουμε όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να δώσουμε ένα κοινό μήνυμα προ όλου του λαού στα Δυτικά Βαλκάνια. Επίση, τα όσα υπόθηκαν, θα ήθελα να σα πω ότι προφανώ το Ηνωμένο Βασίλειο δεν βρίσκεται στο Σέγγεν και τα όσα υπόθηκαν δεν έχουν να κάνουν με μετανάστευση, αλλά με τα ταξίδια. Το σημαντικό είναι να καταφέρουμε να βρούμε μια κοινή βάση με την οποία όλοι να συμφωνούμε. Δεν νομίζω ότι αποκλείουν τόσο πολλοί απόψει μα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε κυρίω για ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν κυρίω με νομική διατύπωση και θεωρώ ότι μπορούμε να γεφυρώσουμε τι ε, διαφορέ μα αυτέ. Ευχαριστούμε η συγκήτρια. Σας ευχαριστώ κύριε Λάτφορτ. Βλέπω ότι όντως κινούμαστε στον ίδιο δρόμο. Θα ήθελα απλώ να τονίσω στο τέλος της συζήτησης αυτής που θεωρώ ήταν ιδιαίτερα επικοδομητική για όλους μας ότι για άλλη μια φορά χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ότι συμφωνούμε και ότι θα καταφέρουμε να ακολουθήσουμε το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχει προβλεφθεί για την ε, κατάργηση υποχρέωσης θεώρησης για το Μαυροβούνιο, τη Σερβία και την Φύρομ και θέλουμε να καταφέρουμε να προωθήσουμε τις ίδιες δυνατότητες και για τη Βοσνία και για την Αλβανία. Με την προϋπόθεση όμως ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να θεωρήσουν ε, ότι η κατάργηση υποχρέωση θεώρηση είναι δεδομένη. Θα πρέπει να συνεχίσουν στον σωστό δρόμο που έχουν ήδη ξεκινήσει, δηλαδή να προσπαθήσουν να ελοποιήσουν τι προποθέσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τι δύο χώρε αυτέ και για του λαού των δύο φτωχωρών. Και για το 25 να σα πω ότι θα πρέπει να βρεθεί και γι' αυτό μια λύση προκειμένου να καλυφθεί, αν θέλετε, αυτό το μαύρο κενό που υπάρχει στα Δυτικά Βαλκάνια. Σα ευχαριστούμε κυρία Φαγιόν, λέει ο Πρόεδρος. Η προθεσμία υποβολής ε, τροπολογιών είναι η 7η Οκτωβρίου και η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας ε, θα γίνει στις 15 Οκτωβρίου. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα τα πράγματα και ότι θα πρέπει μέχρι τότε να βρεθεί μια κοινή συμφωνία μεταξύ όλων των διαφορετικών ε, πλευρών. Σας ευχαριστούμε που θέλουν ε, οι ηγητές να συνεργαστούν με την εισηγήτρια για την συγγραφή της τελικής έκθεσης και θα ήθελα τώρα να περάσουμε στο... Συγγνώμη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να παρέμβει. Παρακαλώ. Θέλετε το λόγο. Ας είστε σύντομοι σας παρακαλώ πολύ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη, λακωνική. Θα ήθελα για άλλη μια φορά να επαναλάβω ότι το ότι προτείναμε μία τροπολογία του κανονισμού 539 για τις ε, χώρες των Βαλκανίων καταδεικνύει για άλλη μια φορά την πολύ μεγάλη πολιτική σημασία που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη γραφική αυτή ζώνη και τη σημασία την οποία δίνουμε για να διατηρήσουμε αυτή την ε, περιφερειακή συνοχή. Όσον αφορά την διαφοροποίηση το ζήτημα αυτό το οποίο έθεσαν κάποιοι ευρωβουλευτές επιτροπή σας όσον αφορά την πρόοδο που είχε σημειώσει η Βοσνία. Το ζήτημα της Βοσνίας δεν έχει να κάνει με την απουσία βιομετρικών διαβατηρίων. Έχει να κάνει με την αξιολόγηση. Η αξιολόγηση θα πρέπει να καλύπτει και άλλους τομείς. Θα πρέπει δηλαδή να δούμε ποια είναι νομοθεσία κατά των διακρίσεων. Το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει δηλαδή να καταλήξουμε σε ένα σύστημα καλύτερης διαχείρισης των συνόρων. Και όλα αυτά εξαρτώνται από προσπάθειες που θα πρέπει να καταβάλει η χώρα και τις οποίες εμείς μέσω αποστολών μας θα πρέπει να επαληθεύσουμε. Δεν πρόκειται για μία αποστολή στην αυτή που θα κάνουμε στο Μαυροβούνιο, στη Σερβία που θα, διαρκέσει μόνο τρεις μέρες. Πρόκειται για μία πολύ πιο σφαιρική αξιολόγηση η οποία θα γίνει τόσο για την Αλβανία όσο και για τη Βοσνία σε σχέση με τα σχόλια της ηγήτριας για τις μικρές αυτές χώρες, τα microstates, τα οποία συζητήσαμε χθε. Θα ήθελα να σας πω ότι εδώ τα πράγματα είναι εντελώ διαφορετικά. Από νομική πλευρά, αυτό που εμεί εντοπίζουμε ω πρόβλημα με την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ότι για μα η τελική απόφαση και η πραγματική κατάργηση υποχρέωση θεώρηση θα πρέπει να γίνει βάση έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το Συμβούλιο ή τους συνομοθέτες στο μέλλον δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για τα μικρά όμως αυτά κράτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στα τέλη του 2006 στο Συμβούλιο μία πρόταση η οποία εγκρίθηκε στη συνέχεια, η αναθεωρημένη δηλαδή πρόταση εγκρίθηκε και τα μικρά αυτά κράτη πέρασαν στο θετικό κατάλογο με την προϋπόθεση βέβαια να υπογραφούν οι κοινοτικέ συμφωνίες απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης. Πρόκειται όμως πάλι για το Συμβούλιο που φασίζει και στην περίπτωση αυτή. Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει τον τελικό λόγο. Βλέπετε λοιπόν πόσο διαφορετικό είναι το νομικό πλαίσιο. Το Συμβούλιο είναι αυτό το οποίο έχει τον τελικό λόγο που φασίζει μετά από πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή μετά από διαπραγμάτευση θα ξεκινήσει με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστούμε. Παρκούν αυτά για τώρα. Λίγοι εδώ ολοκληρώνεται αυτό το σημείο. Περνάμε στο σημείο 18 που αφορά την πρόληψη και διευθέτηση των συγκρούσεων δικαιοδοσίας σε ποινικέ ε, διαδικασίες. Έχουμε το θέμα της έγκρισης ε, του σχεδίου έκθεσης ε, της εισηγήτριας της κυρίας Ρενάτε Βέμπερ. She absent. Απουσιάζει η κυρία Βέμπερ θα λάβει τον λόγο για να την εκπροσωπήσει η κυρία Χανές Πλέσατς, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πρέπει να ζητήσω συγγνώμη για την απουσία της ε, εισηγήτριας κυρίας Ρενάτε Βέμπερ που δεν μπορεί να παραστεί λόγω προβλήματος υγείας εχθές το βράδυ που έπρεπε να πάει στην κλινική. Καλά είναι, αλλά δεν μπορεί να προσέλθει στην Ευρωβουλή σήμερα. Θα προσέλθει αργότερα όταν ε, θα έχει αποκατασταθεί η υγεία της. Υπάρχει συμφωνία ότι τα ευαίσθητα στοιχεία πρέπει με ιδιαίτερη ευαισθησία να αντιμετωπίζονται. Είναι προφανέ αυτό και το γνωρίζουμε αυτό. Θα πρέπει να ανταλλάσσονται μόνο όταν είναι σημαντικά για δίκε σε θέματα ποινική διαδικασία. Αυτό αφορά την ε, απόφαση του ε, Συμβουλίου και αναφέρεται και στο εδάφιο 18 πρώτο τμήμα. Γι' αυτό απόλυτη απαγόρευση όσον αφορά την τροπολογία 2 συμβιβαστική δεν μπορεί να γίνει δεκτή. Θα είμαστε κατά λοιπόν της τροπολογίας 2. Αυτά για να σας ενημερώσουμε πληροφοριακά. Ευχαριστώ. Thank you. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Θα ακούσουμε τώρα από τη Σουηδική Προεδρία τα σχετικά. Η κυρία Ασαβέμπερ. Όχι, δεν θέλετε να παρέμβετε. Δεν θέλετε, εντάξει. Τότε θα ψηφίσουμε για το σχέδιο έκθεσης, εντάξει. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία, έτσι δεν είναι. Χρειάζονται οι κάρτες σας. Να δοκιμάσουμε να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Να δούμε αν λειτουργούν ή όχι οι συσκευέ. Έχετε τι κάρτε σα. we're going to vote. Λοιπόν, θα, κάνουμε, θα ψηφίσουμε το κείμενο. Παράγραφος 5 στα σκεπτικά αιτιολογικές σκέψεις υπέρ χωρίς ηλεκτρονική κάρτα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε μάλιστα αιτιολογική σκέψη 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το 7 όχι θα ελέγξουμε λοιπόν. Λειτουργούν οι συσκευέ. Δεν λειτουργούν τώρα. Λειτουργούν ή όχι. Δεν λειτουργεί. Εντάξει. Can we do? Τι θα κάνουμε, τι θα κάνουμε αν δεν λειτουργούν οι συσκευέ. <laughs> ε? Okay. How many? Πόσοι. Now? Τώρα πόσοι. Δεν λειτουργεί. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας λέγεται στον πρόεδρο να γνωστοποιηθεί. Λοιπόν, η καταμέτρηση θα ψηφίσουμε, αλλά πρέπει να μετρηθούν και εκείνοι που δεν ψήφισαν. Υιοθετήθηκε λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Κύριε Μαστέρα, τι άλλο πρόβλημα. Είμαι αντίθετος. Εντάξει, καταψηφίσατε. και εγώ ήμουν εναντίον. Δεν λειτουργήσε η συσκευή μου. Δύο ψήφοι εναντίον λοιπόν. Και άλλε δύο τι γίνεται. Δύο εναντίον. Τέσσερις λοιπόν εναντίον. Δύο και δύο τέσσερι εναντίον. Δηλαδή 19 ψήφοι εναντίον 29 υπέρ. Υιοθετείται. Υιοθετήθηκε. Αιτιολογική σκέψη 8. Συγγνώμη λέει ο πρόεδρος. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. Αιτιολογική σκέψη 9, τροπολογία 4. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε, τροπολογία 23, είναι ταυτόσιμη λέγεται στον πρόεδρο. Υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. Αποχές, συγγνώμη, αποχές. Καμία αποχή εντάξει εγκρίθηκε. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα πρέπει να ελέγξουμε. Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε για να ελέγξουμε. Παρακαλώ. Τροπολογία λοιπόν 5. Ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα. Ένας από την Άλτε υπερψηφίζουν και δύο από το ΕΛΚ υπερψηφίζουν. Τι γίνεται. Πρέπει να επαναλάβουμε την ψηφοφορία. Επαναλαμβάνουμε την ψηφοφορία. Ξαναρχίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την τροπολογία 5 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Now. Now. The vote is Πέρας ψηφοφορίας. Θα ελέγξουμε. Λέγεται στον πρόεδρο ότι ψηφίζει ένας παραπάνω από το Ψηφίζει ένας παραπάνω που δεν έχει δικαίωμα ψήφου. So it's η τροπολογία αυτή απορρίφθηκε. Συμβιβαστική τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Εντάξει. Λοιπόν, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά αυτή την τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ένας από την άντε παραπάνω ψηφίζει, λέγεται στον πρόεδρο. Θα πρέπει να αφαιρέσουμε έναν από την άντε. Πέρας ψηφοφορίας. have to 25 υπέρ, 26 εναντίον. Αλλά προφανώς φαίνεται ότι ένας από το Άλτε και ένας από το ΕΛΚΑ ψηφίζουν χωρίς να δικαιούνται. Όταν γίνεται ηλεκτρονικός έλεγχος φαίνεται προφανώς ότι υπάρχει ένας από το ΕΛΚ που είναι παραπάνω και ένας παραπάνω από την Άλντε. Συμβαίνει αυτό πράγματι. Τι γίνεται. Πράγματι ούτως έχουν τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει απορρίφθηκε αυτή η τροπολογία. Μάλιστα. Περνάμε στην τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά και πάλι. So. Ψηφίζουμε λοιπόν ηλεκτρονικά την τροπολογία αυτή. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Και τώρα περνάμε στην τροπολογία 24 υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. Απορρίφθηκε μάλιστα. Τώρα η τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. Εγκρίνεται αυτή. Συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Θέλετε να ελέγξουμε κάποιος. Εντάξει, θα ελέγξουμε λοιπόν. Ελέγχουμε και πάλι. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Now the Πέρας ψηφοφορίας τώρα. Εγκρίθηκε επιτέλους αυτή. Τώρα τροπολογία 8. Υπέρ κατά εγκρίθηκε τοπολογία 9 υπέρ κατά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά τέλος ψηφοφορίας εγκρίθηκε Εγκρίθηκε αυτή. Λοιπόν, τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 11. Αποσύρθηκε λέγεται στον πρόεδρο. Γιατί, γιατί όχι την 11. Αποσύρθηκε λέτε μάλιστα. Εντάξει. Η τροπολογία 25 τώρα λοιπόν. Υπέρ. Κατά εγκρίθηκε. Συμβιβαστική τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 12. Όχι, λέτε. Γιατί όχι. Εντάξει, έστω. Πολύ καλά. Ωραία. Τροπολογία λοιπόν 13. Υπέρ. κατά εγκρίθηκε τροπολογία 14 υπέρ κατά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά τροπολογία 14 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε και περνάμε στην τροπολογία 27. Υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε από ό,τι φαίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε η 17 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε η 18 υπέρ κατά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 18 18. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Λοιπόν, απορρίφθηκε. Και τώρα η τροπολογία 29. Υπέρ. Κατά. Φαίνεται ότι απορρίφθηκε. Αυτό είδα. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την τροπολογία 29. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα απορρίφθηκε. Απορρίφθηκε. Λοιπόν, τροπολογία 19 υπέρ κατά εγκρίθηκε τροπολογία 20 υπέρ κατά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 20 άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά τέλος ψηφοφορίας απορρίφθηκε. Τώρα η τροπολογία 21 υπέρ κατά εγκρίθηκε. Τροπολογία 30. 30 έτσι. 30 υπέρ κατά εγκρίθηκε, εγκρίθηκε. Θα κάνουμε τώρα την τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά αυτή τη φορά. Εντάξει, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Σας ευχαριστώ πολύ. Διαδικαστικό, κύριε Μπουσουτήλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να σας προδοποιήσω ότι θέλω να μιλήσω για την τροπολογία 2 και για την τροπολογία 7. Ευχαριστώ πολύ. Okay. Let's proceed. Μάλιστα. Κυρία Κέλλερ, και εσείς διαδικαστικό. Ναι, ναι, για τις τροπολογίε τροπολογίες Επιτροπής Προπολογισμών θα ήθελα διευκρινήσεις για την τροπολογία 2, όπου μιλάμε για τη συνεργασία Frontex και UNHCR στο τελευταίο τμήμα της τροπολογία. τροπολογίας. Δεν είναι σαφές εδώ ποιος θα έχει πρόσβαση στις πληροφορίες ποιου οργανισμού. Τουλάχιστον στη γερμανική εκδοχή φαίνεται ότι η υπηρεσία θα έχει πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες και εφόσον αποφασίσαμε ότι η Frontex δεν θα πρέπει να συμμετέχει στις δραστηριότητες του UNHCR θα πρέπει να συμβαίνει το αντίστροφο, δηλαδή το UNHCR θα πρέπει να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες Frontex. Πρόκειται βέβαια για την ύπατη αρμοστία των για τους πρόσφυγες. Επίσης, στην άλλη τροπολογία είπατε ότι κατά περίπτωση θα ισχύσει. Ξέρω ότι έχουμε εδώ πέρα το κείμενο από τις κατευθύνες γραμμές για τη συνεργασία μεταξύ Frontex και είπα της Αρμοστίας Ηνωμένων Εθνών. Νομίζω ότι η συνεργασία θα πρέπει να γίνεται κατά περίπτωση. Δεν είναι ξεκάθαρο όμως σε ποια περίπτωση αναφερόμαστε εδώ πέρα και ποιος αποφασίζει τελικά. Δηλαδή σε ποια περίπτωση μπορεί η ύπατη αρμοστία να συμμετέχει ή όχι, να συνεργαστεί ή όχι. Ποιος αποφασίζει σε ποια περίπτωση μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο και σε ποια περίπτωση δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Πρόεδρος. Ναι, νομίζω ότι αναφέρεστε εδώ πέρα στην τροπολογία 3 του κυρίου Μπουσουτήλ. Πρέπει να σας κάνω τώρα μια ανακοίνωση. Αν η τροπολογία 3 εγκριθεί, τότε η τροπολογία 2 του κυρίου Ταβάρες και συγκεκριμένα το τμήμα που έχετε εδώ πέρα στα σχόλια θα υποβληθεί στη ψηφοφορία ως επιπρόσθετη τροπολογία με προφορική τροπολογία ουσιαστικά. Ψηφίσουμε την τροπολογία 3, όπως σας είπα, και βάσει το αποτελέσματος της ψηφοφορίας για την τροπολογία 3, στη συνέχεια θα ψηφίσουμε ή δεν θα ψηφίσουμε την τροπολογία 2 του κυρίου Ταβάρες με ένα επιπλέον τμήμα με μια επιπλέον προφορική τροπολογία.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 Κυρία Κέλλερ, να σας δώσω κάποιες διευκρινήσεις για τη γερμανική εκδοχή του κειμένου όσον αφορά την τροπολογία 2 του κυρίου Ταβάρες. Η ε, απόφαση για την ε, συμμετοχή αναπερίπτωση θα γίνει από τα συμβαλώμενα μέρη τα οποία συμμετέχουν σε κάθε επιχείρηση από πλευράς ε, Frontex. Ας προχωρήσουμε σας παρακαλώ στην ψηφοφορία σχέδιο προπολογισμού, σχέδιο έκθεση για τον προπολογισμό. Κυρία Χέντ, διαδικαστικό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λοιπόν, βρίσκω ότι υπάρχει φασαρία στην αίθουσα συζητούν πολύ και δημιουργεί θόρυβο αυτό. Και υπάρχει μεγάλη κίνηση θα έλεγα και ταραχή. Όταν ψηφίζουμε πρέπει να έχουμε ησυχία για να μπορούμε να επικεντρωθούμε στα θέματα στα οποία ψηφίζουμε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ας περάσουμε στην ψηφοφορία. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 3. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Κύριε Μπουσούτιλ, σας ευχαριστώ. Πρωτού ψηφίσουμε την τροπολογία 2, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας πω ότι το ΕΛΚ θέλει να στηρίξει την τροπολογία αυτή με την προϋπόθεση ότι θα είναι επιπρόσθετη ως προς την τροπολογία 3, όπως είπατε κι εσείς, αλλά και αν η τελική διατύπωση case by case basis αντικατασταθούν από το where necessary, δηλαδή το αναπερίπτωση το κατά περίπτωση να αντικατασταθεί από το όπου κρίνεται αναγκαίο, όπου θεωρείται αναγκαίο. Κύριε Ταβάρες. Συμφωνώ ότι όντως πρόκειται για μια επιπλέον τροπολογία, επομένως δεν Υπάρχει εδώ πέρα πρόβλημα με προηγούμενο κείμενο. Θα ήθελα όμω να έχουμε ξεχωριστή, ξεχωριστή ψηφοφορία όσον αφορά την τελευταία διατύπωση, δηλαδή το where necessary. Συμφωνείτε, κύριε Μπουζουτήλ, συμφωνείτε. Ωραία, έτσι θα προχωρήσουμε λοιπόν. Τροπολογία 2 λοιπόν υπέρ. κατά Το ξεκαθαρίσαμε. Ψηφίσουμε αυτή τη στιγμή την τροπολογία με την φράση where necessary, όπου κρίνεται αναγκαίο. where necessary, ε, we're voting Ψηφίζουμε την τροπολογία αυτή τη στιγμή με το where necessary. Κυρία Κέλλερ, διαδικαστικό. Κάνουμε δηλαδή ξεχωριστή ψηφοφορία τώρα και αν δεν εγκριθεί το δεύτερο τμήμα, τότε θα τελειώνει η τροπολογία με τη λέξη activities, δραστηριότητες και τελεία εκεί. Well, and now we're voting on the second part, when necessary. Ψηφίζουμε τώρα το δεύτερο τμήμα where necessary, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4 με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Κύριε Μπουσουτήλ, έχετε ένα διαδικαστικό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Προτού ψηφίσουμε την τροπολογία 7, θα ήθελα να παρουσιάσω μια προφορική τροπολογία με την ακόλουθη διατύπωση. Μετά τον τέλος της Αγγίλης, targeted in general, θα ήθελα να μπει ακόλουθη φράση ή σύμφωνα με υφιστάμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχουν ε, καταρτήσει τα κράτη-μέλη και στη συνέχεια θα συνεχίζεται η παράγραφος ως έχει. Αυτή είναι η προφορική μου τροπολογία. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία αυτή με την προφορική τροπολογία που πρότεινε ο κύριος Μπουσούτιλ. Κύριε Ιακολίνο. Εμείς ε, θέλαμε την τροπολογία Αλφάνο Μπορσελίνο Κροτσέτα. Θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε να την ενσωματώσουμε στο κεφάλαιο που αφορά τις ε, θετικές εμπειρίες ανά το χρόνο, σχετικά δηλαδή με το οργανωμένο έγκλημα. Πώς έχει καταπολεμηθεί στα διάφορα κράτη-μέλη. Εγώ μπορώ να σας δώσω το ιταλικό παράδειγμα το πώς ε, δηλαδή η δικαιοσύνη μπόρεσε να κατασχέσει από για 40 δισεκατομμύρια ευρώ ακίνητα από τους εγκληματίες. Πρόκειται για κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και σκέφτεται να σκεφτόμαστε ότι το να γίνει μία αναφορά στα κράτη-μέλη είναι κάτι το πολύ χρήσιμο για το σύστημα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Μπουσούτη να διαβάσει την προφορική τροποποίηση ώστε να ξέρουμε τι ψηφίζουμε. Μπορείτε να το διαβάσετε παρακαλώ. Shall I do so, Mr. Okay. Να τη διαβάσω πρόεδρε. Εντάξει, ευχαριστώ. Η προτινόμενη προφορική τροποποίηση μετά τις λέξεις στην Αγγίλη θα ξεκινούσαν γενικά και θα ήταν η εξής ή στις υφιστάμενες νομικές διατάξεις και πρωτοβουλίες όπως προτείνονται ή καθορίζονται από τα κράτη-μέλη. Είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Είναι σαφές για όλα τα μέλη τώρα το τι ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Είσουμε το σύνολο του κειμένου τώρα. Υπέρ. Λέγεται στον πρόεδρο να ψηφίσετε ηλεκτρονικά, ηλεκτρονική ψηφοφορία λοιπόν. Περνάμε στην ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. ψηφοφορίας. Yes. Thank you. Σας ευχαριστώ. Υιοθετήθηκε. Ήτανε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

Thank you. Let's Ας συνεχίσουμε, παρακαλώ. Θα ψηφίσουμε τώρα από κοινού κάποιες προτάσεις. Πρόκειται για τις συμφωνίες που συζητήσαμε χθε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αφενός και τον Μαυρίκιο, τον Μπαρμπάντος, τον Άγιο Χριστόφορο Κενέβης, Μπαχάμες, Αντίγκουα και Μπαρμπούντα αφετέρου όσον αφορά την κατάργηση υποχρέωσης θεώρησης. Θα ψηφίσουμε κάθε συμφωνία ξεχωριστά και θα κάνουμε διπλή ψηφοφορία για κάθε συμφωνία. Πρώτα για τη σχέδιο έκθεσης και στο τέλος για το τελικό κείμενο. Γιατί θα κάνουμε τελική ψηφοφορία δηλαδή. Σημείο 20 καταρχάς. Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Μαυρίκιου σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρηση για βραχία διαμονή. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σχέδιο έκθεσης παρακαλώ. Άρκτη ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνεται. Σημείο 21 Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Μπαρμπάντος. Με συγχωρείτε, λέει ο Πρόεδρος. Θα κάνουμε και τελική ψηφοφορία για την προηγούμενη συμφωνία, τελική ψηφοφορία για το σημείο 20, για το Μαυρίκιο δηλαδή. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Σημείο 22 λέει ο πρόεδρος. Σχέδιο έκθεσης πάλι, άρκτη ψηφοφορία. Πέρας. Τελική ψηφοφορία τώρα για την ίδια έκθεση. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Σας ευχαριστώ. Εγκρίνεται. Σημείο 23. Μπαχάμες. Σχέδιο έκθεσης πάλι ψηφίζουμε αυτή τη στιγμή. Άρθρη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τελική ψηφοφορία για την ίδια έκθεση άρθρη ψηφοφορία. Πέρας. Σας ευχαριστώ. Εγκρίνεται. Σημείο 24. Αντίγκουα και Μπαρμπούντα. Ψηφίζουμε το σχέδιο έκθεσης, άκτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται και τελική ψηφοφορία για την ίδια έκθεση, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Πολύ ωραία. Το σύνολο τώρα των προτάσεων αυτών έχει εγκριθεί. Α, ξεχάσαμε τις Σεϊχέλες. Δεν το είδα, λέει ο Πρόεδρος. Δεν έφτασα μέχρι τις Σεϊχέλες, σας ζητώ συγγνώμη. Άρτη ψηφοφορία για το σχέδιο έκθεσης. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τελική ψηφοφορία για την ίδια έκθεση, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή, τον κύριο Μπουζουτήλ. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας στην ψηφοφορία. Και έχουμε τώρα το σημείο 26. Σαν Κίτσε Νέβης, Άγιος Χριστόφορος και Νέβης, μα ψηφίσαμε για την έκθεση αυτή. Νομίζω ότι ψηφίσαμε το σύνολο των προτάσεων. Σεχέλες, Μπαρμπάντος, Ξεχάσαμε να ψηφίσουμε το σημείο 22. Πολύ ωραία. Ας επιστρέψουμε στο σημείο 22. Άγιος Χριστόφορος και Νέβης ψηφίζουμε το σχέδιο έκθεσης άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Και τελική ψηφοφορία για την ίδια έκθεση. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα πραγματικά σας λέω με βεβαιότητα ότι εγκρίθηκαν όλες οι προτάσεις, όλες οι προτάσεις, όλες οι εκθέσεις του κυρίου Μπουζουτήλ. Ας Περνάμε στο σημείο 26. Κοινή συζήτηση με τα μέλη της Υποεπιτροπής για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι μια ανταλλαγή απόψεων με τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Θεμελιωδών, ε, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Καλωσορίζουμε πρώτα τα μέλη της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την πρόεδρο της Υποεπιτροπής κυρία Χαουταλά. Επίσης ε, τον κύριο Μόρτεν Κέρον προσκεκλημένο μας, ε, Διευθυντή της Υπηρεσίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον οποίο η δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή έχει στενές σχέσεις. Προτείνω να υπάρξουν εναλλάξε ερωτήσει μεταξύ των μελών και των ε, ε, φιλοξενουμένων. Κάποιοι όμως ανήκουν και στις δύο επιτροπές. Η κυρία Χάταλα, την οποία καλωσορίζουμε, θα προεδρεύσει σε αυτό το τμήμα της ανταλλαγής ε, απόψεων. Πριν όμως θα δώσουμε τον λόγο στον κύριο Μόρτεν Κιέρομ για μια σύντομη εισήγηση, εισαγωγή. Θα θέλαμε λοιπόν να ακούσουμε την εισαγωγή του κυρίου Κιόραμ από πλευρά της Υπηρεσίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Και για μας όσοι είμαστε νέα μέλη της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, ΛΥΜΠΕ, θα είναι επικοδομητικό και θα μας βοηθήσει να αξιολογήσουμε τη συνεισφορά της υπηρεσίας αυτής για την προπαρασκευή του προγράμματος της ημερήσιας διάταξης της Στοχόλμης. Ο κύριος Μόρτεν Τσέρομ λοιπόν έχει πρώτος τον λόγο. Καλώς ήρθατε βέβαια, έχετε εσείς πρώτος τον λόγο και μετά θα ακούσουμε την κυρία Χάταλα. Παρακαλώ. Ο κύριος Τσέρομ. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σας ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε να προσφωνήσω εσάς σε αυτή την κοινή συζήτηση σήμερα εδώ. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μένα που μπορώ να σας προσφωνήσω όλους σας σε αυτή τη φάση ενωρίς της θητείας, της κοινοβουλευτικής σας και προσβλέπω στη συνεργασία αναμεταξύ μας στα επόμενα πέντε χρόνια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ήταν πάντα υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την πρώτη κοινή διακήρυξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων το 1977 σε εκατοντάδες προτάσεις ψηφίσματος διάφορες διαφορετικές γενναίες ευρωβουλευτών, κοινοβουλευτικών εκπροσώπων εξέφρασαν ανησυχίες για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε χώρες μακριά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε χώρες που βρίσκονται μέσα στις 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν προκλήσεις όχι μόνο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εντός. Και αυτό είναι το μέλημα, κύριο μέλημα της ε, Υπηρεσίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Να αναφέρω κάποια μόνο. Ρατσισμός και ξενοφοβία, <clears throat> μισαλοδοξία, Ισλαμοφοβία, κοινωνικός αποκλεισμός των τσιγκάνων, των Ρωμά, αύξηση όσον αφορά την καταγραφή των ανταλλαγών προσωπικών δεδομένων, ομοφιλοφιλοφοβία, αρνητικές διακριτικές, ε, αρνητική διακριτική μεταχείριση σε, μειονεκτικά άτομα, σε άτομα με μειονεξίες ε, όσον αφορά όσους έχουν AIDS, κακοποίηση παιδιών κτλ. Αυτά είναι μόνο λίγα, λίγες από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και όλα αυτά τα θέματα πραγματικά συμβαίνουν και καλύπτονται στο πολιετές αυτό πλαίσιο για την υπηρεσία μας. Πολιετές πλαίσιο που ξεκίνησε και φτάνει ως το 2012 και που θα υλοποιήσουμε την εντολή μας μέσα στο πλαίσιο αυτών των θεμάτων και αυτών των εντολών. Σε πολλά από αυτά τα θέματα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη προσφέρει κάποιες λύσεις νομοθετικά με την πολιτική της, με χρηματοοικονομικά μέσα κτλ. Από τα ευρωβαρόμετρα και τα ερωτηματολόγια γνωρίζουμε ότι τρεις από τους τέσσερις Ευρωπαίους θέλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίζει μεγαλύτερο ρόλο και να επηρεάζει περισσότερο τα πράγματα όσον αφορά την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για να υλοποιηθούν όμως αυτές οι προσδοκίες, η αποτελεσματικότητα της ανταπόκρισης στις μεγάλες αυτές προκλήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενδυναμωθεί. Εσείς ως συνομοθέτες και ως αρμόδια αρχή για τον προϋπολογισμό στα δημοσιονομικά θα διαδραματίσετε κύριο ρόλο επ' αυτών. Ας στραφώ τώρα στην εντολή της υπηρεσίας μας. Τι κάνουμε δηλαδή σχετικά. Είμαστε ακόμα μια νέα, νεαρή υπηρεσία που θεσπίστηκε τον Μάρτιο 2007 συγκροτήθηκε και είμαστε μία από τις πιο μικρές από τις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που μπορούμε να σας προσφέρουμε είναι τρία πράγματα. Πρώτον, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούμε να προσφέρουμε συγκριτικά στοιχεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων που εντάσσονται μέσα στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να αξιολογήσετε τις επιπτώσεις και τα κενά, τα χάσματα που υπάρχουν. Δεύτερον, μια ανεξάρτητη πραγματογνωμοσύνη όσον αφορά συγκεκριμένα προβλήματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να ταυτοποιήσετε τις ανάγκες για δράση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν τέλει, να δώσουμε ένα εργαλείο, ένα μέσο για να υπάρξει συνειδητοποίηση μεταξύ των Ευρωπαίων για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και οι καλύτερες νομικές διατάξεις έχουν μικρό αποτέλεσμα αν η συνειδητοποίηση για το πώς μπορεί να διεκδικήσει κανείς αυτά τα δικαιώματα απουσιάζει υπηρεσία μπορεί να είναι καταλήτης για αυτή τη μεγαλύτερη συνειδητοποίηση. Έτσι λοιπόν, εν συνόψη, πρέπει να, δώσουμε, να δίνουμε γνωμοδότηση και πραγματογνωμοσύνη τεκμηριωμένη στα ευρωπαϊκά όργανα για τα θέματα που αφορούν ε, <clears throat> τους Ευρωπαίους πολίτες και αφορούν τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η πρόσθετη αξία ποια είναι. Είναι η επικέντρωση στα κενά και χάσματα που υπάρχουν όσον αφορά την υλοποίηση των στόχων για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ενώ είναι σημαντικό να υπάρχουν προδιαγραφές, από την άλλη πλευρά αντιμετωπίζουμε πρόβλημα και ελλείψεις στην υλοποίηση και εκτέλεση. Εδώ λοιπόν η Ευρωπαϊκή αυτή υπηρεσία μπορεί να διαδραματίσει ένα ρόλο, ένα ρόλο κλειδιού για να δείξει πού βρίσκονται κενά και πώς πρέπει να καλυφθούν. Για παράδειγμα, είδαμε ότι σε σχέση με την μη διακριτική μεταχείριση και την ομοθεσία είδαμε ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν μπορούν να αναζωογονηθούν και να διασφαλιστούν μόνο με νομικές προβλέψεις και κατοχυρώσεις. Έχουμε και μια τεράστια ε, επισκόπηση που έγινε όσον αφορά εθνικές μειονότητες και τους μετανάστες. EU Mides. Αυτό το EU Mides ερωτηματολόγιο όσον αφορά χιλιάδες άτομα από τις μειονότητες στα 27 κράτη-μέλη και τα στοιχεία αυτά τα οποία δείχνουν ότι αντιμετωπίζουν αρνητική διακριτική μεταχείριση, ρατσιστική μεταχείριση. Η πλήρης έκθεση θα παρουσιαστεί εφέτος το Δεκέμβριο σε εκδήλωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Βλέπουμε ότι υπάρχουν υψηλά επίπεδα εξακολουθούσας διακριτικής αρνητικής μεταχείρισης και ρατσισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν καταγράφονται και δεν αναφέρονται. Για παράδειγμα, ένας σε δύο τσιγκάνους ζει και βιώνει αρνητική διακριτική μεταχείριση. Βίωσε τέτοια μεταχείριση στους τελευταίους 12 μήνες, το τελευταίο έτος. 11 τέτοια συμβάντα ανά έτος κατά μέσο όρο. Και πρέπει να λάβουμε επιπλέον υπόψη ότι μόνο μια πολύ μικρή μειονότητα μειοψηφία αυτών των ατόμων αναφέρουν και καταγγέλουν τις περιπτώσεις αρνητικής μεταχείρισης στις αρχές. Είτε είναι η αστυνομία αυτές οι αρχές, είτε άλλη αρχή. ένα παρόμοιο πρότυπο απέρευσε και από την έκθεσή μας για την ομοφυλοφοβία στα κράτη-μέλη. Και πάλι εδώ η αρνητική διακριτική μεταχείριση δεν αναφέρεται και δεν καταγγέλλεται, δεν καταγράφεται από τι αρμόδιε αρχέ. Η έκθεση για την ομοφυλοφοβία ε, συντάχθηκε μετά από αίτημα τη Ευρωβουλή. Το EU Mides και η έκθεση για την ομοφιλοφοβία αποκαλύπτουν εκπληκτικά χαμηλά επίπεδα ε, σε γνώση αυτών των πραγμάτων όσον αφορά τα άτομα μειονοτήτων όσον αφορά τα μέσα για να προστατευτούν και να διεκδικήσουν δικαιώματα και να προστατευτούν έναντι ρατσιστικών επιθέσεων. Τέσσερα από πέντε άτομα δεν γνωρίζουν καμιά οργάνωση ή οργανισμό που μπορούν να τους δώσουν υποστήριξη σε τέτοια συμβάντα. Έτσι δεν στρέφονται λοιπόν ούτε στην αστυνομία, ούτε στα θεσμικά όργανα τα οποία δημιουργήθηκαν για να τους προστατεύουν. Αυτά τα στοιχεία υπογραμμίζουν και τονίζουν στους πολιτικούς στα κράτη-μέλη ότι περισσότερα κονδύλια πρέπει να επενδυθούν για να υπάρξει αύξηση της συνειδητοποίησης και ευαισθητοποίησης και όσον αφορά και την υλοποίηση και διεκδίκηση των δικαιωμάτων αυτών των ατόμων. Υπό το φως λοιπόν Τη έρευνα τη Υπηρεσία για τα θεμελιώδη δικαιώματα πρόσφατα είχαμε την ευκαιρία από τη Σουηδική Προεδρία που μας την προσέφερε αυτή την ευκαιρία να σχολιάσουμε για το μελλοντικό πρόγραμμα της ημερήσια διάταξης τη Στοχόλμη. και ξέρω ότι θα το συζητήσετε το απόγευμα αυτό. Έχει καθοριστεί αυτή η ημερήσια διάταξη για το μέλλον τη Ευρώπη στον τομέα τη δικαιοσύνη και των εσωτερικών υποθέσεων αυτοί οι τομείς φυσικά έχουν την πιο άμεση επίπτωση για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι θετικό ότι η Μελλοντική Επιτροπή έχει δεσμευτεί να δώσει μεγαλύτερα κίνητρα και να αναλάβει πρωτοβουλίες για την διάσταση για τα ανθρώπικα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης ελπίζουμε ότι θα υλοποιηθεί υπό τον κανονισμό των διατάξεων της Λισαβόνας, της συνθήκης Λισαβόνας, που θα κάνει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα θεμελιώδη δικαιώματα πολύ πιο ευδιάκριτα ό,τι μέχρι σήμερα. Δεσμευτική χάρτα για τα θεμελιώδη δικαιώματα μέσω της συνθήκης, η πρόσβαση και της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σύμβαση, για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η, η προσυπογραφή κατά της αρνητικής διακριτικής μεταχείρισης, θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων υπογραμμίζουν την δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ των μειονοτήτων. Μέσα στο πλαίσιο όλων αυτών των νέων νομικών θα έλεγα διατάξεων και δομών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα είναι μόνο αναγκαίο, θα είναι φυσικό να ενταχθούν φυσιολογικά και φυσικά τα θεμελιώδη δικαιώματα σε όλο το νομοθετικό έργο και την ομολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλωσορίζουμε το γεγονός ότι η Ευρωβουλή αρκετές φορές έχει ζητήσει ο ρόλος αυτός της υπηρεσίας να λαμβάνεται υπόψη όταν προτείνεται σχετική νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να εντάσσονται οι πτυχές για τα ανθρώπινα δικαιώματα θεμελιώδη δικαιώματα. Θέλω να τονίσω ότι η υπηρεσία μας έχει πολύ στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους στην σκηνή και στο επίπεδο των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δεν είμαστε οι μόνοι εμπλεκόμενοι, ιδιαίτερα το Συμβούλιο της Ευρώπης και στο εθνικό επίπεδο οι εθνικοί οργανισμοί και θεσμοί για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αντίστοιχοι αξιωματούχοι ε, των κυβερνήσεων για αυτή την ε, δραστηριότητα. Επίσης έχουμε και το, την, Euro, ε, Frontex, την Europol, την Eurojust και φυσικά και το Ίδρυμα για την Ισότητα των Φύλων. Αυτό που χρειαζόμαστε ως Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν θα θεωρεί την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων ως ένα εγχείρημα διοικητικό ή διακυβέρνησης, αλλά που θα το εξετάζει σε βάθος για να είναι σεβαστή σεβαστά τα δικαιώματα αυτά. Μια ειδική υπηρεσία μπορεί να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να εντάξει αυτές τις πτυχές των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλες τις πολιτικές της Ένωσης, εμπνέοντας έτσι, δίνοντας πνεύμα και ψυχή στην θεμελιώδη χάρτα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη ζωή όλων των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ειλικρινής μου ελπίδα ότι οι δύο κοινοβουλευτικές σας επιτροπές θα συνεχίσουν να είναι η αιχμή του δόρατος σε αυτή τη διαδικασία. Μπορώ να σας διασφαλίσω ότι είμαστε στη διάθεσή σας για να σας υποβοηθήσουμε με τα αναγκαία στοιχεία και τεκμήρια ώστε να τεθούν στο επίκεντρο της διάταξη διάταξης Ευρωπαϊκής Ένωσης τα θεμελιώδη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Με χαρά θα δούμε να μας επισκέπτεστε στην έδρα μας στη Βιέννη κάποτε μελλοντικά. Ευχαριστώ. So, ευχαριστούμε. Θα πάρει τώρα το λόγο η κυρία Χαουτέλα και στη συνέχεια ευρωβουλευτές άλλοι έχουν ζητήσει τον λόγο και μπορούμε να κάνουμε και συζήτηση συνέχεια. Κυρία Χαουτέλα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μας δίνετε τη δυνατότητα να έχουμε την κοινή αυτή συνεδρίαση με μέλη δηλαδή της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο κύριος Κέρουμ είχε πάρει το λόγο στο παρελθόν και ενώπιον της δικής μας Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και εκ μέρους της δικής μου επιτροπής θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό που είπατε, ότι δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει μια ευθυγράμμιση της εφαρμογής των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι στα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλο και περισσότερο τα θεμελιώδη δικαιώματα και όχι μόνο βέβαια σε εξωτερικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να βελτιώσει τα αποτελέσματά της για τα θεμελιώδη δικαιώματα στο εσωτερικό της προκειμένου να γίνει πιο πιστική όταν προσπαθεί να παραδειγματίσει τρίτες χώρες, ιδίως στα πλαίσια συμφωνιών εμπορικών συναλλαγών. Και επίσης να σας θέσω ένα ακόμα ερώτημα. Πιστεύετε ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι τομείς ανησυχίας, δηλαδή τομείς ε, για τους οποίους ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση επεκρίνεται από τρίτες χώρες ότι δεν ακολουθεί δηλαδή τα ίδια τα δικά της κριτήρια για την ε, τήρηση και την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και θα ήθελα να σας ζητήσω να έρθετε και στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όταν θα συνεδριάσουμε αργότερα αυτό το μήνα στο Στρασβούργο με μέλη της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Θα ήταν πολύ σημαντική η παρουσία σας σε μια τέτοια συνεδρίαση γιατί ε, ε, ουσιαστικά οι ειδικέ αρμοδιότητε συνάδουν πάρα πολύ με τι αρμοδιότητε Επιτροπή αυτή, αλλά βέβαια και με τι αρμοδιότητε Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, στην οποία βρισκόμαστε σήμερα. Πολύ ωραία. Χάνε Πλάσα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Χάουταλα που ήρθατε, ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Σίγουρα έχουν γίνει πρόοδοι σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά λείπουν πολλά ε, ακόμα να γίνουν σε πρακτικό επίπεδο. Έχετε την αίσθηση ότι η Κομισιόν χρησιμοποιεί όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της ούτω ώστε να πιέσει τα κράτη-μέλη να σεβαστούν τις υποχρεώσεις του για τα θεμελιώδη δικαιώματα εγώ πιστεύω ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο και πρέπει να χρησιμοποιούμε τη διαδικασία παραβίασης όταν πρόκειται για παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να ξέρω τη γνώμη σας επ' αυτού. Μιλήσατε επίσης για μία έκθεση ε, και η Κομισιόν ερωτήθη σχετικά ε, πριν από λίγο καιρό. Τώρα, δεδομένων των προβλημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έπρεπε η έκθεση να συντάσσεται κάθε χρόνο. Η Κομισιόν θεωρεί ότι είναι πολύ καλή ιδέα. Δεν θεωρείτε κι εσείς ότι πρέπει να γίνεται σε αιτήσια βάση αυτή η έκθεση. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ που ήταν και σύντομος. Σύντομη, με συγχωρείτε. γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε την πρωινή μας συνεδρίαση στις 12.30. Και υπάρχουν αρκετοί ακόμα συνάδελφοι που θέλουν το λόγο, επομένως σας παρακαλώ πολύ να περιοριστείτε, να περιορίσετε τις παρεμβάσεις σε δύο μόνο λεπτά, κυρία Καλ. Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση άκουσα τον ε, Διευθυντή της Υπηρεσίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και ως πρώην εισηγήτρια για την υπηρεσία αυτή. Είχα δώσει πραγματικές μάχες προκειμένου να δημιουργηθεί, να υλοποιηθεί το σχέδιο της υπηρεσίας αυτής. Και χαίρομαι πραγματικά που βλέπω ότι ε, γνωρίζουν πλέον πώς να εργάζονται, πώς να συνεργάζονται με τις υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες και την Ευρωπαϊκή Ένωση Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη με τα πορίσματα της υπηρεσίας αυτής και ιδιαίτερα με το προσωπικό έργο του Διευθυντή της Υπηρεσίας. Ωστόσο, έχω ένα πρόβλημα. Πώς όλο το ζήτημα των διακρίσεων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων θα πρέπει να τα διαχειριστούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πιο συγκεκριμένα στην υπηρεσία. Θέτω λοιπόν το ζήτημα αυτό γιατί θα προκύπτει όλο και περισσότερο και κάθε μέρα βλέπουμε ότι ανακύπτει το ζήτημα αυτό και ότι έχουμε τελικά δύο μέτρα και δύο σταθμά. Έχουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις διάκρισης, περιπτώσεις πάρα πολύ σημαντικές και σοβαρές. Έχουμε εκθέσεις, έχουμε ψηφίσματα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Και συμφωνώ με αυτά που είπαν και οι συνάδελφοι ότι θα πρέπει να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς όλες τις περιπτώσεις ε, αρνητικής διάκρισης. Θα υπήρχαν όμως και άλλες περιπτώσεις που θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε, περιπτώσεις που θεωρούνται όμως ευαίσθητες και τελικά δεν τις προσεγγίσουμε ποτέ, δεν ασχολούμαστε ποτέ μαζί τους και τελικά δεν επιλύουμε τα προβλήματα αυτά. Αναφερθήκατε στις μειονότητες, πολύ πρόσφατα εγκρίναμε σχετική νομοθεσία στην, ε, ε, για μια περίπτωση διακριτικών μεταχειρήσεων στην Σλοβακία, όπου υπήρχε διακριτική μεταχείριση κατά μειονοτήτων. Ε, πρόκειται για έκδηλη διάκριση κατά των μειονοτήτων και δεν έγινε τίποτα στην περίπτωση αυτή, μόνο ότι υπάρχουν κοινοτικέ νομοθεσίε κατά των διακρίσεων. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω ποια είναι η δική σα άποψη γιατί πολλοί πολίτες πιστεύουν πλέον ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι η κατάσταση. Έχει έρθει πλέον η ώρα να πούμε ότι σαφώς υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις διακρίσεων, θα πρέπει όμως να τυχαίνουν τις ίδιες μεταχείρισεις στο ίδιο επίπεδο. Πάνω από 20 ευρωβουλευτέ θέλουν το λόγο και έχουμε με το ζόρι 20 λεπτά μπροστά μα. Παρακαλώ πολύ λοιπόν να είστε πολύ σύντομοι στις παρεμβάσει σα. Και κλείνω κατάλογο των ομιλητών επίση, η κυρία Φλότχα. Ε, ευχαριστώ. Κυρία και κύριε συμπρόεδροι, με μεγάλη χαρά εμείς πάντοτε παρακολουθούμε τους απολογισμούς σας γιατί εμείς ε, χρειαζόμαστε ακριβώς την ανεξάρτητη πραγματογνωμοσύνη την οποία συντάσσεται και μας βοηθάτε μας τους νομοθέτες να βελτιώνουμε τις προδιαγραφές των ευρωπαϊκών πολιτικών. Το χρειαζόμαστε αυτό στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης που είναι πάρα πολύ σημαντικό και που αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της ε, Στοκχόλμης. Ρωτώ, οι τροπολογίες που προτείνατε για την προστασία και αλληλεγγύη προβλέπουν ε, εργασίες και προτάσεις και εισηγήσει που θα μπορούσατε εσείς να υποβάλλετε για τις προτάσεις επανεισδοχής ε, η πανεισδοχή δημιουργεί συνήθως ε, προβλήματα παρανομίας ε, για τους μετανάστες. Ή οδηγούν σε προβλήματα με τους ετούντες ασύλου. Υπάρχουν άνθρωποι που προτιμάνε να κόψουν το δάχτυλό τους για να μην τους πάρουν τα δαχτυλικά αποτυπώματα για να τα βάλουν στην Eurodac. Λοιπόν, τι λέτε εσείς για όλα αυτά. Έχετε ωραία νέα να μας αναγγείλετε για το μέλλον. Η κυρία Στανόκα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συνεχίσω τα όσα είπε η πριν από λίγο συνάδελφο για μια διαφορετική προσέγγιση που θα πρέπει να υπάρχει τα εξωτερικά προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτός δηλαδή Ευρωπαϊκή Ένωση και εντό Ευρωπαϊκής Ένωση. Αν συγκρίνεται εκθέσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα από το παρελθόν, κάθε φορά που αναφερόμαστε για τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωση, ακολουθούμε άλλη στάση, ενώ όταν μιλάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Κατάνιο νομίζω ότι είχε κάνει μια τέτοια έκθεση, δεν αναφερόμαστε σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη, ενώ κατονομάζουμε τρίτες χώρες πολύ εύκολα, δεν κατονομάζουμε ποτέ κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν, υπάρχουν, όταν υπάρχει παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και κύριε Κέρουμ, θα ήθελα να συνεχίσουμε τη συζήτηση που ξεκινήσαμε πριν από λίγο. Πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε ένα τέτοιο πρόβλημα. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις ε, αναφορές που υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εσείς μας είπατε ότι δεν είναι εκεί σας αρμοδιότητα να ασχοληθείτε με τις αναφορές αυτές. Αλλά, για παράδειγμα, τον Απρίλιο ασχοληθήκαμε με μία έκθεση, με μία αναφορά που είχε υποβληθεί κατά το παρελθόν έτος και όχι μόνο μία αναφορά μάλλον, πάρα πολλές ε, αναφορές με συγχωρείτε είχαν να κάνουν με παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η δική σας υπηρεσία θα μπορούσε να εξετάσει τις αναφορές αυτές και να μας βοηθήσει με την εμπειρογνωμοσύνη που έχει σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστούμε ο κύριος Μωράης. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Γκάλ και ε, Στανόκα αναφέρθηκαν και στο ζήτημα αυτό για τις αποφάσεις που μπορούσαν να ληφθούν και για τις γνωμοδοτήσεις που εσείς μπορείτε να κάνετε. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πολύ συχνά ανακύπτει και στις συζητήσεις που γίνονται στην Ολομέλεια. Θα ήθελα να θέσω ένα βασικό ερώτημα, κάτι στο οποίο αναφερθήκατε στην αρχή της παρουσίασής σας. Έχουμε διατάξεις κατά των διακρίσεων στον χώρο εργασία, για παράδειγμα, οι οποίε όμω ισχύουν, υποτίθεται από το 2000. Θα πρέπει όμω όλα τα κράτη-μέλη να αρχίσουν να εφαρμόζουν την νομοθεσία αυτή και θα πρέπει η νομοθεσία αυτή πλέον να περάσει στη βασική νομοθεσία όλων των κρατών μελών. Αναφερθήκατε σε εθνικές αρχές και υπηρεσίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα κράτη-μέλη στην εφαρμογή των νομοθεσιών αυτών. Δεν υπάρχουν όμως τέτοιες αρχές και υπηρεσίε σε πάρα πολλά κράτη-μέλη. Τι μπορεί λοιπόν να γίνει για αυτό το έλλειμμα εφαρμογής της κοινοτική νομοθεσίας. Τι μπορείτε εσείς να κάνετε σαν υπηρεσία προκειμένου να βοηθήσετε ή να υποχρεώσετε τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν μια κοινοτική νομοθεσία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσημα έχει τη διαδικασία επιπαραβάση. Δεν λειτουργεί όμως πάντα η διαδικασία δεν λειτουργει ομω παντα η διαδικασια αυτη Πάρα πολλά κράτη επικαλούνται την αρχή τη επικουρικότητα προκειμένου να μην εφαρμόσουν τι κοινοτικέ διατάξει κατά των διακρίσεων. Εσεί ω υπηρεσία θεμελιωδών δικαιωμάτων τι μπορείτε να κάνετε. Ευχαριστούμε κύριο Βανχέκ. Κύριε Κλάις, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριος Φαν Χέκε είναι συνάδελφος σε άλλη όμως κοινοβουλευτική επιτροπή. Λοιπόν, ο κύριος Διευθυντής είναι ανάμεσά μας. Γι' αυτό θέλω να δραχθώ τις ευκαιρίες να κάνω κάποιες παρατηρήσεις για τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι ετήσιες εκθέσεις ε, από την Υπηρεσία για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα συντάσσονται. Παρακολουθώ τα τεκτενόμενα με αυτή την υπηρεσία εδώ και κάποια χρόνια και πώς συντάσσονται οι εκθέσεις. Και πάντα διατυπώνω το ερώτημα, δεν θα ήταν δυνατόν έννοιες όπως ρατσισμός και αρνητική διακριτική μεταχείριση να καθοριστούν, να προσδιοριστούν σε στενότερο πλαίσιο πιο εξειδικευμένα. Στην τελευταία έκθεση για το ρατσισμό και την αρνητική μεταχείριση βλέπω κάποιες περιπτώσεις να αναφέρονται που σε, σε κάποια σχολεία, σε κάποια κράτη-μέλη απαγορεύονται οι μαντήλες, οι κεφαλομαντήλες ή οποιαδήποτε κάλυψη της κεφαλής. Υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι Υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι που δεν συσχετίζονται με το ρατσισμό για την απαγόρευση αυτή. Σε αυτήν όμως την ετήσια έκθεση αναφέρεται σαν να ήταν τεράστιο πρόβλημα αυτό που αφορά τον ρατσισμό και την αρνητική διακριτική μεταχείριση. Ενώ δεν συμβαίνει πάντα κάτι τέτοιο. Γι' αυτό θα ήθελα να απευθύνω έκκληση. Τέτοιου είδους περιπτώσεις και πράγματα πιο σύνετα και πιο προσεκτικά να τα αντιμετωπίζετε. Να μην δημιουργείται εντύπωση ότι ισοπεδώνονται όλα και αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο χωρίς να ανήκουν στο ρατσισμό και στην αρνητική μεταχείριση. Ευχαριστώ κύριο Σπόβο. Σε ευχαριστώ πολύ. Η κυρία προηγούμενα το ανέφερε και εγώ. Πρέπει να τονίσω από πλευράς μου και πάλι ότι στη Ρουμανία μας ανησυχεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι εξτρεμιστικές δυνάμεις στη Ρουμανία και με τον ε, γλωσσικό νόμο της Σλοβακίας όπως είδαμε και σε σχέση με το κόλλημα το οποίο ε, βίωσε ο πρόεδρος του κράτους σε σχέση με τη Σλοβακία βλέπουμε συμβάντα παρόμοια με εκείνα της Σλοβακίας. Συνάδελφοι ανέφεραν πράγματα που και εγώ θα ήθελα να τονίσω. Απομένει μια ερώτηση που θέλω να διατυπώσω. Δεν θεωρείτε ότι τα παλαιά και τα νέα κράτη-μέλη όταν έρχεται η στιγμή να γίνει λόγος για τις παραβάσεις και παραβιάσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, όταν πρόκειται ακριβώς και θέλουμε και να εξετάσουμε νομοθετήματα και νόμους που προστατεύουν εθνοτικές μειονότητες, τους τσιγκάνους από την αρνητική διακριτική μεταχείριση, να έχουμε μια κοινή επικέντρωση. Και έτσι αν συνέβαινε κάτι τέτοιο δεν χρειαζόταν εσείς να συντάσετε να συντάσσετε εκτενείς εκθέσεις για παραβιάσεις και παραβάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πώς μπορεί λοιπόν να προωθηθεί η υπόθεση αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση διότι εμείς στην τελευταία κοινοβουλευτική θητεία δώσαμε αυτή την προώθηση, υπογραμμίσαμε αυτή την ιδέα, δυστυχώς όμως μας παρακόλλησαν οι, οι ηγέτες των δύο μεγάλων πολιτικών ομάδων να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Και η ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχουν μια κοινή συνεδρίαση. Μία παρατήρηση, μία ερώτηση εσείς ε, απαριθμήσατε διάφορες ευρωπαϊκές υπηρεσίες ε, με τις οποίες συνεργάζεστε. Δεν βρήκα το Ίδρυμα του Δουβλίνου για την βελτίωση των ε, συνθήκων εργασιακής εργασίας και θα ήθελα να το αναφέρω αυτό για την έρευνα και για τις επαφές σε σχέση με τις τοπικές αρχές και τις κοινότητες μεταναστών ε, και στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και δυτικών κρατών και ανατολικών κρατών ε, καθότι γνωρίζω. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η έρευνα λοιπόν. Και το δεύτερο θέμα αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα τα ίδια εκτός όμως Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η ερώτηση που είναι όσον αφορά για μας τον πιο ε, κοντινό μας ε, γείτονα και που βρίσκεται στην ανατολική γειτονία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι όμως μία από τις τελευταίες ευρωπαϊκές χώρες όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι σεβαστά, όπου συλλαμβάνονται οι πολίτες για πολιτική δράση που έχουν και επίσημα αναγνωρίζονται αυτά τα άτομα ως ε, κρατούμενη συνείδησης Amnesty International και αυτό νομίζω θα πρέπει να ληφθεί από εσάς υπόψη σε σχέση με το έργο σας. Thank Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ντερόκα παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας, κύριε. Κυρίως όσον αφορά τους τσιγκάνους και που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα αυτό και πολύ σημαντικά τα στοιχεία που έχετε αναφέρει. Μία από τι ερωτήσει που θα ήθελα να θέσω είναι ακολουθώντα τον κύριο Μόραη και την ερώτησή του. Εκπλήσω με πράγματι μαθαίνοντα ότι όταν έρχεται η στιγμή εφαρμογή των οδηγιών και στην τελευταία έρευνα αναφέρεται ότι υπάρχει διαχωρισμό εθνοτικό στις περισσότερε πρώην κομμουνιστικές χώρες ε, στην Ευρώπη. Θα ήθελα να ξέρω σε ποιο βαθμό Ίδια ερώτηση δηλαδή του κυρίου Μωράης. Τι γίνεται σε σχέση με τα, τους πόρους που χρειάζονται για να καταπολεμήσουμε αυτά τα συμβάντα, διότι έχουμε σημαντικές παραβιάσεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και η άλλη πτυχή είναι όσον αφορά την οικονομική κρίση. Σε ποιο βαθμό είναι το Ίδρυμά σας, ο φορέας σας ε, σε θέση να κατανοήσει το τι προκαλεί η οικονομική αυτή κρίση μεταξύ των διαφορετικών ε, κοινωνικών και εθνοτικών ομάδων. Κατά πόσον έχετε προχωρήσει όσον αφορά αυτό. Ευχαριστώ. Okay, Mr. σας ευχαριστώ κύριος Τόκας παρακαλώ. Igazgató gratulálok Πρέπει να ευχαριστήσω και εγώ τον Γενικό Διευθυντή της Υπηρεσίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Τον συγχαίρω. Επίσης ε, και σε σχέση με την κυρία Κιγκακάλ, Επίσης ε, η συγχαρητήρια διότι υπήρξε η δημιουργία αυτής της πολύ σημαντικής υπηρεσίας. Διότι εγώ εκείνο από το γεγονός ως αφετηρία, όπως είπε και η κυρία Χάουλα, ότι εμείς πολλές φορές στρεφόμαστε στα προβλήματα τρίτων χωρών περισσότερο έντονα και δεν στρεφόμαστε με τον ίδιο τρόπο έντονα στα δικά μας προβλήματα. Ξεχνάμε και αμελούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των μειονοτήτων και των δικαιωμάτων τους και των ελέγχων μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε δύο μέτρα και σταθμά. Είναι πολύ πιο εύκολο να κάνει λόγο, λόγο κανείς για τους Ουιγούρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωβουλή αντί για τους Τσάγκος ε, στην Ρουμανία ή τους Ούγγρους, στη Σλοβακία. Πρέπει να αλλάξει αυτή η κατάσταση πια. Τα θρησκευτικά δικαιώματα, τα γλωσσικά δικαιώματα, τα δικαιώματα των μειονοτήτων είναι πάρα πολύ σημαντικά πεδία. Όπως για παράδειγμα τα δικαιώματα των Ούγγρων που ζουν στην Σλοβακία, στην Ρουμανία. Εκείνοι κατά τη διάρκεια θρησκευτικών τελετών δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ίδια τη μητρική τους γλώσσα. Δεν μπορούν να ακούσουν το κήρυγμα του κληρικού, του παπά στην ίδια τη λειτουργία, στην μητρική τους γλώσσα. Χρειαζόμαστε λοιπόν σίγουρα έναν ομπουσμαν Ευρωπαίο που θα προστατεύει τα μειονοτικά δικαιώματα αυτών των μειονοτήτων. Χρειαζόμαστε ένα αξίωμα, μια τέτοια αρχή ή φορέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. ευχαριστώ. Um, Λυπούμε που έχασα την έναρξη αυτή τη πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση λόγω του ότι είχαν λυμμένε υποχρεώσει σε άλλη κοινοβουλευτική επιτροπή. Θα ήθελα να ξέρω αν η κρίση για τα ανθρώπινα δικαιώματα που αφορά την Ουγγαρία, που συνεχίζεται για τρία χρόνια τώρα, έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη εργασιών τη υπηρεσία σα. Γνωρίζετε ότι το 2006, το φθινόπωρο του 2006, υπήρξαν ε, βιαιότητες, μαζικές αστυνομικές βιαιότητες ε, και χτυπήθηκαν πάμπολα άτομα ε, ξεκίνησαν αβάσιμες αστήρικτες ε, κατηγορίες ε, και ένα από τα γεγονότα ήταν ότι το κόμμα Φίδες σε μια συνάντηση τώρα έχουμε και εκπρόσωπο τις φίδες, ε, την κυρία Κίνγκο Γκάς, ε, που σίγουρα μπορεί σε σχέση με, αυτά τα, με αυτές τις περιπτώσεις ε, να αποσαφηνίσει τα πράγματα. Αυτή ήταν η αφετηρία τότε. Τα τελευταία τρία χρόνια από τότε τα πολιτικά και <clears throat> ανθρώπινα δικαιώματα στην Ουγγαρία παραβιάζονται και σε μεγάλο βαθμό και αυτό είναι κάτι το σίγουρα απαράδεκτο. Σε σχέση με τον Ombudsman στην Ουγγαρία διαπιστώθηκε με βάση δεκάδες δικαστικές αποφάσεις από το Ανεξάρτητο Συμβούλιο Παραπώνων εις βάρος της αστυνομίας. Η υπηρεσία σας θα έλεγα δεν θα ήταν αξιόπιστη αν αυτή την υπόθεση και κλείνατε τα μάτια όσον αφορά και τις παραβιάσεις αυτές που είναι κατάφορες των ε, ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ένα κράτος μέλος από την Ανατολική Ευρώπη πρέπει να ντρέπονται ότι ένα μέλος της κυβέρνησης της ε, Ουγγαρίας τότε που ήταν μέλος της κυβέρνησης όταν έγιναν οι μαζικές βιαιότητες από την αστυνομία με διαταγή της κυβέρνησης ένα μέλος αυτής της τότε κυβέρνησης είναι μέλος της Επιτροπής LIBE στην Ευρωβουλή και απευθύνω έκκληση στους ψηφοφόρους και στους πολίτες της Ευρώπης να υψώσουν τη φωνή τους εναντίον αυτού του έσχους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Γενικέ Διευθυντά, θα ήθελα να σας καλωσορίσω εδώ στην δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή και να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία να σας ακούσουμε. Χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό, επειδή είναι και η πρώτη μου φορά στην Ευρωβουλή, η πρώτη μου θητεία και η ερώτησή μου συνδέεται με τα οικονομικά κοινωνικά θέματα και την κρίση που είχε επίπτωση σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η, Ευρωπαϊκή, η υπηρεσία σας έκανε μια ανάλυση για το πώς αυτή η κρίση είχε επιπτώσεις και επηρέασε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ποιε είναι οι διαφορέ και τι συμβαίνει σε σχέση με τα διαφορετικά κράτη-μέλη. Ένα άλλο θέμα είναι. Στην έκθεσή σα, εσεί αναφέρετε και λέτε ότι οι πολίτες δεν έχουν συνειδητοποιήσει και δεν γνωρίζουν σε ποια θεσμικά όργανα μπορούν να στραφούν όταν έχουμε παραβιάσεις ε, και παραβάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τέσσερις από τους πέντε πολίτες, είπατε, δεν γνωρίζουν την ύπαρξη τέτοιων θεσμικών οργάνων και οργανισμών. Πώς θα έπρεπε να διαχέεται η πληροφόρηση αυτή ώστε να ε, ε, συνειδητοποιούν και να ευαισθητοποιούνται οι πολίτες. Διότι όταν υφίστανται κάτι οι πολίτε δεν γνωρίζουν σε ποιον να στραφούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τζέρομ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. πως έχω μπροστά μου μισή ώρα, <laughs> μπορώ να μιλήσω. Πρέπει να αστομεύετε. Είναι 12.30 ώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω συνοπτικά στις περισσότερες ερωτήσεις. Ακούστηκαν κάποιες παρατηρήσεις που είχαν να κάνουν με την εξωτερική και εσωτερική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς ως υπηρεσία ασχολούμεθα μόνο με τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχουμε αρμοδιότητα, δεν έχουμε εντολή για τις εξωτερικές σχέσεις. Τούτου λεχθέντος βέβαια, όπως είπε και η πρόεδρος κυρία Χάουταλα, υπάρχει μια άμεση συσχέτιση ανάμεσα στο τι κάνουν τα 27 κράτη-μέλη στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς αντικατοπτρίζεται αυτό εξωτερικά, στις σχέσεις δηλαδή που έχουν με τρίτες χώρες. Απαντώντας λοιπόν στην ερώτησή σας θα έλεγα ότι ένας από τους τομείς όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη έχουν πολλά να προσφέρουν στις εξωτερικές τους σχέσεις, αλλά υπάρχει και περιθώριο βελτίωσης, είναι πρώτον να αποδεχθούμε ότι υπάρχουν προβλήματα αν δούμε διάφορες περιοχές στις τρίτες χώρες θα συνειδητοποιήσουμε ότι δεν υπάρχει αναγνώριση συγκεκριμένων προβλημάτων και να πούμε ότι όχι μόνο να γνωρίζουμε τα προβλήματα αλλά ότι καταβάλουμε προσπάθειες για να τα αντιμετωπίσουμε, για να τα επιλύσουμε, ότι έχουμε τις κατάλληλες αρχές και τα θεσμικά όργανα τα οποία μας επιτρέπουν σε κοινοτικό επίπεδο να ξεπεράσουμε τα προβλήματα αυτά. Όχι μόνο τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και το Συμβούλιο της Ευρώπης, για παράδειγμα. Κατά αυτόν τον τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα η Ευρώπη θα καταφέρει να δώσει μια πιο ενωμένη εικόνα προς τα έξω. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν αυτό το, αυτά τα θετικά χαρακτηριστικά που έχουμε. Μια άλλη ομάδα ζητημάτων έχει να κάνει με αυτό που ανέφερα πριν από λίγο, δηλαδή με, την εφαρμογή, με την, το έλλειμμα εφαρμογής της νομοθεσίας. Υφίσταται δηλαδή νομοθεσία, αλλά σαφώς υπάρχουν και κάποια νομοθετικά κενά ακόμα, δεν έχουμε καλύψει τα πάντα, αλλά υπάρχει και ένα ζήτημα προβλήματος εφαρμογής νομοθεσίας και η υπηρεσία είναι μοναδική στο ότι είναι η μόνη υπηρεσία που έχει πλέον την εντολή να εξετάσει πραγματικά το πρόβλημα του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της ισλαμοφοβίας, των αρνητικών διακρίσεων κατά τον Ρώμα. Εμείς μπορούμε πλέον να εξετάσουμε με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια τα προβλήματα αυτά που ταλανίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και δεκαετίες. Να δούμε ακριβώς τι γίνεται από πλευράς ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. και να δούμε το πρόβλημα του, το, ότι υπάρχει μία απουσία θέλετε καταγγελιών προς τις αρμόδιες αρχές, προς την αστυνομία, ότι όλες αυτές οι περιπτώσεις ρατσισμού για παράδειγμα δεν καταγγέλλονται. Και ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε με την γνώση αυτή όχι μόνο να ενημερώσουμε εσά, αλλά θα καταφέρουμε να ενημερώσουμε και τα απαραίτητα όργανα, τους απαραίτητους φορείς προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και τις αστυνομικές αρχές, και εργαζόμαστε εδώ πέρα με τη ΣΥΠΟΛ και με άλλους φορείς, θα μπορέσουμε δηλαδή μέσω της συνεργασίας αυτής να καταρρύψουμε τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν όχι μόνο για τις εθνοτικές μειονότητες, αλλά γενικότερα για τους πολίτες εκείνους οι οποίοι πέφτουν θύματα αρνητικής διαχείρισης λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού ή για άλλους λόγους. Ελπίζουμε λοιπόν ότι η καλύτερη αυτή δυνατότητα που θα έχουμε εξέταση των προβλημάτων αυτών και η γνώση που θα αποκομίσουμε θα χρησιμοποιηθεί όχι μόνο από εμά αλλά και από άλλους αρμόδιους φορείς και θα πρέπει να καταφέρουμε να έχουμε και μια καλύτερη μεθοδολογία για να κάνουμε έρευνε και θα πρέπει να εμπνευστούν από τη μεθοδολογία αυτή και τα κράτη-μέλη. Γιατί α το αποδεχθούμε στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν γνωρίζουμε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε διάφορε υπρεσιονιστικέ, θα έλεγα, νομοθεσίε που εγκρίνονται, όπου έχουμε απλώ μια γενικότερη αίσθηση ότι κάτι δεν πηγαίνει πολύ καλά. Με την γνώση που θα καταφέρουμε να αποκομίσουμε, νομίζω ότι θα καταφέρουμε να νομοθετούμε και πιο συγκεκριμένα στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τώρα τι μειονότητε, αυτό είναι ένα άλλο ξεχωριστό ζήτημα. Σαφώς δεν κάνουμε ε, διάκριση για το ποιος πέφτει θύμα διάκρισης ή όχι και για ποιους λόγους. Επομένως ασχολούμεθα σαφώς και με τις εθνοτικές μειονότητες και μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επεξεργαζόμαστε τώρα μια έκθεση ακριβώς για τις μειονότητες. και εφόσον εγκριθεί η συνθήκη της Λισαβόνα, θα δημιουργηθεί μια καλύτερη διασύνδεση ανάμεσα στις εθνοτικές μειονότητες και την ε, υφιστάμενη νομοθεσία προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μια, ένα σχετισμό που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει καλύτερα η υπηρεσία μας για να προστατεύσει τις μειονότητες. Κάτι ακόμα και ολοκληρώνω. Ετέθησαν πολλές ερωτήσεις που είχαν να κάνουν με την οικονομική κρίση. Εμείς συστήσαμε μια ομάδα εργασίας στην υπηρεσία μας που ονομάζεται RADAR που έχει ως στόχο να καταφέρει να εξετάσει σφαιρικά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκειμένου να γνωρίζουμε ακριβώς ποιε είναι οι επιπτώσεις τη οικονομική κρίση, χρησιμοποιώντας διάφορες παραμέτρους το όλο εγχείρημα τελικά φάνηκε να είναι πιο πολύπλοκο από ό,τι είχαμε φανταστεί στην αρχή. Αποκομίσαμε όμω πολλά διδάγματα και θα προσπαθήσουμε τώρα να επεξεργαστούμε καλύτερα τα διδάγματα αυτά και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήσαμε. Και στον τομέα αυτό συνεργαζόμαστε με τη Frontex, γιατί και αυτοί έχουν ανάλογου μηχανισμού προκειμένου να είναι σε θέση να ενημερώνονται για τα ζητήματα αυτά. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε μια ανησυχητική επίπτωση οικονομικής κρίσης δεν προκαλεί εντύπωση ότι ε, ορισμένα από τα άτομα που απολύθηκαν πρώτα ήταν άτομα που προέρχονται από μειονότητες. Μία μικρή ομάδα από αυτούς ενδεχομένως να επέστρεψε στην χώρα προέλευσής τους, στη χώρα καταγωγή τους. Οι υπόλοιποι πιστεύω ότι θα πέρασαν στην παράνομη αγορά ή σε αυτό που ονομάζουν ε, μερικοί ευρωπαϊκή αγορά δουλείας, δηλαδή κατάφορη εκμετάλλευση ουσιαστικά. Καταλαβαίνετε ότι για την υπηρεσία μας είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταφέρει να διεισδύσει στο πρόβλημα αυτό. Το εξετάζουμε πάντως και προσπαθούμε να δούμε πώς θα καταφέρουμε να το εντάξουμε και αυτό στο πρόγραμμα εργασίας μας. Αυτά είχα να σας πω σε μια πρώτη φάση κύριε Πρόεδρε. Ολοκληρώνω λοιπόν στο σημείο αυτό και προσβλέπω πραγματικά στον ε, συνεχή διάλογο και συνεργασία που ε, θέλω να έχω με τη δική σας Επιτροπή. Εξ ονόματος και των δύο Επιτροπών θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ θερμά κύριε Πρόεδρε για την εξαιρετική σας παρουσίαση και φυσικά για την ότι ύπαρξη αυτής της υπηρεσίας για τα θεμελιώδη δικαιώματα που είναι ένα επίτευγμα που παγκόσμια μπορούμε να είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ και οι δύο κοινοβουλευτικές επιτροπές θα είναι σε επαφή μαζί σας κύριε. Και έχω την εξή ε, ανακοίνωση και οι δύο επιτροπές μας θα συνέλθουν στις 15.00 στις 3 το απόγευμα σε αυτή την αίθουσα πάλι. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ κύριε Λόπεθ Αγγιλάρ για αυτή τη συνεργασία.